Mm. Good morning. Um, we have to start. Καλημέρα σας. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε. Στις 11 και 4 θα έρθει ο Υπουργός Υγείας της Βουλγαρίας. Οπότε ας ξεκινήσουμε για να προλάβουμε. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να δώσουμε το λόγο στον συγκεκριμένο τον κύριο Λαβία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή εισαγωγή στα πλαίσια της σημερινής συζήτησης και γιατί εντάξαμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη, γιατί νομίζω ότι η νομοθετική πλαισίωση έχει μεγάλη σημασία για να ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου και ε, τα προνόμια μας. Θα υποβάλω και ορισμένα ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΜΑ που είναι παρούσες για να έχουμε διασαφήσεις και εγγύησεις. Θα ήθελα να σας πω πώς έχουν καταρχήν τα πράγματα, γιατί η ΕΜΑ που βρίσκεται στο Λονδίνο θα πρέπει να μεταφερθεί μέχρι τις 30 Μαρτίου 2019 από το Λονδίνο αλλού, γιατί είναι η ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις 22 Ιουνίου του 2017 οι επικεφαλής των 27 ενέκριναν μία ειδική διαδικασία για, την, ε, για τη μεταφορά αυτή. Και στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών Γενικών Υποθέσεων της 20ης Νοεμβρίου του 2017 αποφασίστηκε ε, η μεταφορά όλων των οργανισμών που είχαν έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η αίμα θα, μεταβεί, θα πάει στο Άμστερνταμ. Πρόκειται για μια διαδικασία που προβλέφθηκε και όπως ξέρετε δύο ήταν οι προτινόμενες ε, έδρες. Στις 29 Νοεμβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για να γίνει η μεταφορά της αίμα από το Λονδίνο στην Ολλανδία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έλαβε πληροφορίες καθόλου ως προς τη διαδικασία. Μέχρι ότου μετά τη διαδικασία μάθαμε ότι η όλη διαδικασία δεν βασίζεται στις συνθήκες αλλά σε μια κοινή δήλωση των αποκεντρωμένων οργανισμών που είναι μια πράξη μη δεσμευτική νομικά. Εν ώψη αυτής της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να επικρίνω την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής της ε, νέας έδρας της ΕΜΑ. Και όπως σας είπα πριν έγινε κλήρωση. Ε, μη λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της απόφασης έγινε λόγος για μια διαδικασία η οποία ήταν συνοπτική. Και στην ουσία τι έγινε, έγινε μια υποτυπώδης κλήρωση σαν να παίζαμε χαρτιά. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο, σημαντικές, δύο σημαντικούς οργανισμούς που έχουν επίπτωση στη ζωή των πολιτών, όπως είναι η αίμα. Κάτι το οποίο έχει σημασία για τον έλεγχο της ασφάλειας των φαρμακευτικών σκευασμάτων για ανθρώπινη χρήση. Θεωρώ λοιπόν ότι οι διαδικασίες που ε, ακολουθήθηκαν δεν έγιναν, ε, δεν γνωστοποιήθηκαν μάλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δύο αυτές περιπτώσεις. Και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορέσαμε να συμμετάσχουμε στις διαδικασίες επιλογής της έδρας των ευρωπαϊκών οργανισμών. Με την εφαρμογή της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας, της συναπόφασης, όπως προβλέπεται από τις συνθήκες. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προβάλλει τα προνόμια και τις εξουσίες του, τροποποιώντας αν το κρίνεται σκόπιμο ένα μέρος της απόφασης της Κομισιόν έτσι ώστε να έχουμε πλήρη και αποτελεσματική εργασία της ΕΜΑ χωρίς διασπάθηση του δημοσίου χρήματος για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους που εκπροσωπούμε εδώ. Δεν είναι καθόλου δημοκρατικό το ότι αποκλείστηκαν οι πολίτες από αποφάσεις τέτοιου τύπου. Ε, λήφθη μια απόφαση που δεν είναι νομικά δεσμευτική και δεν ενεπλάκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε πληροφοριακά για να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες πρωτίστως, με βάση τις οποίες έχουμε δικαίωμα συναπόφασης. Και νομίζω ότι αν συμφωνήσουν οι άλλες πολιτικές ομάδες θα πρέπει να προσαρτήσουμε μία πολιτική δήλωση υποτύπων joint statement για να ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία. Έχω λοιπόν μία σειρά ερωτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για να τηρήσουμε τη διαδικασία που θα μας οδηγήσει στην οριστική ε, μεταφορά της έδρας μετά το Brexit. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν η Επιτροπή μας επιβεβαιώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πλήρεις εξουσίες στα πλαίσια αυτής της ε, κανονιστικής ε, διαδικασίας. Άρα οι κοινέ δηλώσεις δεν έχουν νομική ισχύ. Και το ρωτώ γιατί στο ανακοιναθέν τύπου μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται το πλήρες ανακοινωθέν και στην ουσία ε, εφαρμόζονται οι νέες έδρες των δύο οργανισμών, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο το οποίο επιβεβαιώνει τέτοιες επιλογές. Και στην ουσία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να επιβεβαιώσει αποφάσεις άλλων, κάτι το οποίο δεν μου φαίνεται καθόλου σωστό. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο ελέγχει τη διαδικασία που θα μας οδηγήσει στη μεταφορά της έδρας της ΕΜΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και να μας πει σε ποιο σημείο βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες έτσι ώστε να δούμε τι θα κάνουμε με την προσωρινή έδρα της, ε, του ίδιου του οργανισμού και κατά πόσο μπορεί να μας εγγυηθεί ότι η μεταφορά θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι τις 30 Μαρτίου του 2019, μέσα στα πλαίσια της ε, σωστής και χρηστής λειτουργίας του οργανισμού καθίσταται σαφές ότι θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τι μπορεί να μας πει για τις εργασίες ε, για το Vivaldi Building, δηλαδή την τελική έδρα του ΕΜΑ. Ποια είναι, ποιο είναι το χρονικό διάστημα που προβλέπετε για την έδρα αυτή και πότε θα είναι έτοιμη για να υποδεχτεί τον οργανισμό φαρμάκων και αυτό με βάση τελική διατύπωση που προβλέπετε. Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης κατά πόσο αυτή η διπλή μεταφορά στην ουσία πλήττει τη λειτουργία του οργανισμού και κατά πόσο μπορεί να μας εγγυηθεί για την σωστή συνέχεια των εργασιών μετά το Μάρτιο του 2019. Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια κοινή ερώτηση προς την Επιτροπή και την ΕΜΑ σε σχέση με την προσωρινή έδρα. Κατά πόσο θεωρούν και οι δύο, η Επιτροπή και η ΕΜΑ, ότι οι χώροι που είναι διαθέσιμοι, οι χώροι υποδοχής εμπειρογνωμόνων μπορούν να εγγυηθούν τη σωστή λειτουργία, ενδιάμεση λειτουργία, προσωρινή λειτουργία της, ε, του οργανισμού. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θα υπάρχει διπλό κόστος μεταφοράς, δηλαδή από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ και κατά πόσο θα πρέπει να ενταχθεί στο κόστος του Brexit δηλαδή θα καταβληθεί το κόστος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η δεύτερη όμως μεταφορά, αυτή που θα γίνει μεταξύ προσωρινής έδρας και ε, η μεταφορά στο Άμστερνταμ, στο Vivaldi Building, από ποιον θα καλυφθεί, από την Ολλανδία θα ήθελα να υπάρχουν εγγυήσεις από την Επιτροπή ότι δεν θα εγγραφεί ούτε ένα ευρώ στον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Γιατί δεν ε, συμβαδίζει με τις αρχικές προδιαγραφές. Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω την ΕΜΑ ποιες είναι οι συνέπειες στην περίπτωση διακοπής διαπραγματεύσεων για το Brexit ή εάν προτρέξουμε στη συμφωνία ως προς την τελική προθεσμία, 30 Μαρτίου δηλαδή του 2019. Η αίμα θα μπορέσει να μεταφερθεί προγενέστερα αν αποφασιστεί με βάση αυτά που ακούσαμε και εχτές για μια μεταβατική περίοδο του Brexit. Αυτά μας είπε ο βασικός διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μίλησε για μια μεταβατική περίοδο εξόδου όπου θα ισχύει ένα status quo. Σε αυτή την περίπτωση η μεταφορά του οργανισμού θα πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως γιατί στις 30 Μαρτίου του 19 θα χάσει ο οργανισμός ορισμένα προνόμια και ιδιαίτερα το προσωπικό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσο σε αυτή την περίπτωση θεωρεί η Επιτροπή ότι αυτή είναι η ημερομηνία όπου όλα θα πρέπει να είναι ε, έτοιμα για τη μεταφορά. Τελευταία ερώτηση προς την ΕΜΑ. Εάν υπάρξει προγενέστερη συμφωνία, θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει μία μεταφορά πριν από τις 30 Μαρτίου του 19 ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Λαβία, για το σχέδιο έκθεσης και για τη δουλειά που έκανε. Η έκθεση και γενικώ η όλη διαδικασία πρέπει να οργανωθούν πολύ σωστά για να μην δημιουργηθεί οποιαδήποτε ανασφάλεια και για να τηρήσουμε και τις προθεσμίες. Γιατί εδώ μιλούμε για τη ζωή των πολιτών των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικογένειές τους ε, και οι ίδιοι πρέπει να έχουν ε, την απαραίτητη πληροφόρηση και μια σωστή διαδικασία για να μπορέσουν να οργανώσουν τη ζωή τους και την, με την κατάστασή τους. Συμφωνώ με αυτά που λέει ο κύριος Λαβία για την όλη διαδικασία. Και πιστεύω ότι αυτή θα πρέπει να είναι η τελευταία φορά που το Κοινοβούλιο αποφασίζει με τέτοιο τρόπο, που τίθεται προ Η κοινή, η κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων το 2012, όταν το Κοινοβούλιο παραιτήθηκε του ρόλου του για να επιλέξει την έδρα, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να τεθεί ε, ως δεδομένο και θα πρέπει να μπει και στην ε, ημερήσια διάταξη για συζήτηση και χαίρομαι που οι συνάδελφοι από την ΑΦΚΟ έχουν συμπεριληφθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα για τις δύο αυτές φάσεις της μετεγκατάστασης της υπηρεσίας του οργανισμού θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες ότι οι φορολογούμενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα χρειαστεί να δαπανίσουν ούτε ένα λεπτό παραπάνω για τη μετακατάσταση αυτή και τις δύο φάσεις. Και επίσης, ε, ο οργανισμός από τον προπολογισμό του σίγουρα δεν θα μπορέσει να καλύψει όλο το κόστος της μετακατάστασης Η χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης θα πρέπει να υπάρξει και αυτό αναφέρεται και στο εισαγωγικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά καλό θα ήταν ίσως να μπει και σε κάποια αιτιολογική σκέψη. Επίσης θεωρώ ότι είναι καλό να συμφωνήσουμε για την έδρα της, ε, του οργανισμού και να υπάρξει ένα λεπτομερές πλαίσιο το οποίο θα την ε, καλύπτει για τη χώρα που θα τη φιλοξενεί. Η Κομισιόν στη δήλωσή τη λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει πριν από την ίδια την μεταγκατάσταση, αλλά νομίζω ότι αυτό παρά είναι ασαφέ και μπορεί να δημιουργήσει κάποια ασάφεια. Οπότε ε, ο εκπρόσωπο του οργανισμού θα πρέπει να μα το σχολιάσει. Και όπως και ο εισηγητής, έχω και εγώ κάποιες αμφιβολίες. Η Κομισιόν θα μπορούσε ή ο οργανισμός να μας πούν τι γίνεται σε περίπτωση, με τη μετακατάσταση σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο ε, αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν το τέλος του Μαρτίου 2019 ή αν ε, παγώσουν οι διαπραγματεύσεις, αν καταρρεύσουν. Και επίσης να ρωτήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον οργανισμό να μας πούν εάν η Ολλανδική κυβέρνηση ε, πληρεί τις υποχρεώσεις που τις έχουν τεθεί και αν προχωρούν τα πράγματα όπως έχουν σχεδιαστεί ή αν υπάρχει χώρος ή ανάγκη για βελτίωση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να σας θυμίσω ότι έχουμε λίγο αυστηρόχρονο διάγραμμα. Η κυρία Κρούπα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητού. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε έτσι όπως έχουμε σχεδιάσει. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην τύχη για την επιλογή της ε, έδρας ενός τόσο σημαντικού οργανισμού. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομη θα είμαι, κυρία γιατί ξέρει πολύ καλά ο εισηγητή ότι συμφωνώ με τη θέση του και με τα ερωτηματικά που θέτει και τον ευχαριστώ που οργάνωσε μια συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα με τους σκιώδεις εισηγητέ στο Στρασβούργο. Είναι σύντομη η έκθεση του, η, γνωμοδότησή του, αλλά υπενθυμίζει τα ουσιαστικά την ε, μετακίνηση του οργανισμού και το θέμα του κόστους. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αναλάβει το κόστος τη μεταφορά και μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Brexit. Και επειδή θα υπάρξει καθυστέρηση της πράδοσης του κτηρίου Βιβάλντι, νομίζω ότι οι κάτω χώρε θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος της προσωρινής λύσης. Όπως ε, είπε και ο σοσιαλιστής ε, εισηγητής, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε το κόστος αυτό να βαρύνει τον προπολογισμό της Ένωση. ούτε το ένα κόστο ούτε το άλλο. Τώρα, κάποια βασικά θέματα για το μέλλον. Εδώ ως ε, κοινοβούλιο τίθενται κάποια θέματα διαδικασίας και δεν θέλουμε κι εμεί ε, να επηρεαστούμε από πράγματα εξωτερικά. Ε, επίσης, η διαδικασία, επαναλαμβάνω, η διαδικασία του Συμβουλίου ξεκίνησε με μια κλήρωση στην, με μια ε, πραγματικότητα. Αυτό τι σημαίνει, ότι καταπίπτει κάθε επιχειρηματολογία. Τουλάχιστον στο γαλλόφωνο τύπο, ε, αυτό έβγαλε έναν απόϊχο ως μια ε, τύπου επιπλέον αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αυτή τη διαθεσμική συμφωνία, υποτίθεται από το 2012 και είναι η βάση όλων αυτών και στην πραγματικότητα μας κλέβει το προνόμιο να συνεισφέρουμε στις επιλογές. Ξέρουμε τη σημασία της έδρας του οργανισμού. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε αυτές τις επιλογές. Αυτή η κοινή δήλωση του 2012 θα πρέπει να την καταγγείλουμε Στι συζητήσεις μας στο Στρασβούργο, ο εισηγητή ξέρει πολύ καλά ότι ήμουν λιγάκι πιο ρίζοσπαστική. Προφανώς συμφωνώ να συνοδεύσουμε το κείμενό μας με μία δήλωση που είναι ουσιαστική. Για να πούμε ότι είναι η τελευταία φορά. Τελεία. Δεν θα το ξαναδεχτούμε. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρουμε θέση. Ξέρουμε βεβαίω ε, παράλληλα ότι δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ριζοσπαστικοί. Υπάρχουν θέματα υγεία εδώ. Υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα τα οποία εμπλέκονται. Δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε τη διαπραγμάτευση, δεν μπορούμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, όμως θέλουμε να μας ακούσουν. Θέλουμε να δούμε όλοι μαζί με ποιον τρόπο θα συνοδεύσουμε αυτή τη ε, δήλωση, με ποια λόγια θα την τύσουμε, ούτω ώστε να είμαστε αξιόπιστοι και να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Διαβάζοντα το κείμενο του εισηγητή, ε, θέλω να σα κάνω μια πρώτη πρόταση. Διαβάζοντα το άρθρο 2 που εκφράζει την κατάπληξή μα για, τα, το πώς διενέθησαν τα πράγματα. Το Κοινοβούλιο, η, διαδικασία θα πρέπει να περάσει στην ε, τακτική νομοθετική διαδικασία. Θα πρέπει, πρέπει να πούμε, να περάσει στην συνήθινη νομοθετική διαδικασία καλύτερα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα κάνουμε το κείμενο λιγάκι πιο έντονο. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, λέει η κυρία Κονέτσκα, Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Λαβία, ο οποίος στην εισαγωγική του δήλωση έθεσε κάποια ερωτήματα, τα οποία παραμένουν απάντητα για όλους μας. Και αφορούν κυρίως το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων με αυτή την κίνηση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει τροχοπέδι στη λειτουργία του. Όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές, διαφωνώ που το Κοινοβούλιο στην γνωμοδότησή ε, του προτείνει αλλαγές στην ε, επιλογή της έδρας. Πιστεύω ότι είναι εντελώ ε, ανεύθυνο για τους υπαλλήλους του οργανισμού που αρχίζουν να προγραμματίζουν τη νέα του ζωή στο Άμστερνταμ. Η διαδικασία για την επιλογή της έδρας δεν ήταν ιδανική. Η τελική απόφαση βασίστηκε σε λοταρία ουσιαστικά. Ρίξαν το νόμισμα, πούμε, και, κεφαλή γράμματα. Κορώνει γράμματα. Καταλαβαίνω γιατί επιλέγει συγκεκριμένη έδρα, ε, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι ένα κεντρί ε, για τα κεντροευρωπαϊκά κράτη που τους είχαν υποσχεθεί πιο ενδιαφέρουσες agencies, πιο ενδιαφέροντες οργανισμούς και ποτέ τους, τους δώσανε. Εάν ποτέ το θέμα ε, τεθεί ως πολιτικό ερώτημα, νομίζω ε, ότι θα βλάψει τελικά το Κοινοβούλιο και θα δημιουργήσει αρνητική εικόνα. Εκεί που θα πρέπει να μπει πιο δυνατά το Κοινοβούλιο είναι στο θέμα της διαδικασίας, όπως για, για τον συγκεκριμένο οργανισμό, την, τον ΕΦΣΑ και άλλους οργανισμούς, είναι απαράδεκτη. Κάποιες βασικές ε, υπηρεσίες, κάποιοι βασικοί οργανισμοί που είναι επίσης ε, σημαντικοί για την υγεία μας και την προστασία της υγείας μας υποχρηματοδοτούνται και δεν μπορούν να κάνουν τις μελέτες τους, θα πρέπει να βασίζονται στα αποτελέσματα άλλων και το γεγονός ότι αυτό είναι προβληματικό το έχουμε δει και έχει αποδειχθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω να υποσκάψω την σημερινή συζήτηση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε σε θέματα πολύ σημαντικά για το μέλλον των οργανισμών αυτών. Ευχαριστώ, κυρία Όκεν. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να συζητήσουμε περισσότερο την εντολή του οργανισμού. Ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Το θέμα της α, ανεξαρτησίας του. Και όχι αυτά που συζητάμε εδώ. Δυστυχώς είμαστε εγκλωβισμένοι λιγάκι στη συζήτηση γύρω από την έκθεση Λαβία. Βεβαίω, συμφωνώ με τον κύριο Λαβία με κάποιε αποχρώσει διαφορετικέ, ε, τι οποίε άκουσα από άλλου ομιλητέ, αλλά γενικά συμφωνώ ε, με αυτόν. Με συγχωρείτε, αλλά το κορώνα ή γράμματα, α πούμε, είναι ότι πιο γελίο υπάρχει σε επίπεδο διαδικασία. Τι είναι αυτά. Τότε να οργανώσουμε έτσι μια λοταρία για οτιδήποτε, α πούμε. Λαχιοφόρο αγορά θα. Και με λαχιοφόρο αγορά θα αποφασίζουμε τα πάντα. Ε, μιλάμε τώρα για γελιότητε, παραλογισμού και γελιότητες. Και επίσης είναι επώδυνο να συμβαίνει κάτι τέτοιο ε, μέσα σε απόλυτη αδιαφάνεια χωρίς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν ήδη. Θέλω να κλείσω με δύο πράγματα. Πολλοί ομιλητέ είπαν να σκεφτούμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το Στρασβούργο ως διαπραγματευτικό χαρτί για να αποφύγουμε ας πούμε το περιφερόμενο τσίρκο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακόμα μια φορά. Εάν αποφασίσουμε να μην επιλέξουμε κάτι τέτοιο, ε, το επιλέγουμε γιατί δεν είναι πρακτικό να πηγαίνουμε στο Στρασβούργο. Το αεροδρόμιο δεν είναι καθόλου πρακτικό. Και δεν είναι και εύκολο για μας να μετακινούμαστε. Ίσως να το εξηγήσουμε. Να εξηγήσουμε γιατί έχουμε τέτοια προβλήματα. Να εξηγήσουμε ότι έχουμε προβλήματα με τις μεταφορές. Για να το καταλάβει και ο κόσμος. Επίσης, θα πρέπει τη δεύτερη μετακίνηση του οργανισμού ε, να την πληρώσουν η, η, Ολλανδία, οι κάτω χώρες και να μην κοστίσει ούτε ένα σεντ στον κοινωτικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Λαβία, λέει η κυρία Σρέζερ Πιέρη. Εδώ μιλάμε για εργαζόμενους και για δημόσια υγεία ουσιαστικά, μιλώντας για αυτόν τον οργανισμό. Στις κάτω χώρε, μας άρεσε το, ο τρόπος με τον οποίο αποφασίστηκε να μετακινηθεί ο οργανισμός. Μας αρέσει η απόφαση επίσης. Και το γεγονός ότι οι δύο οργανισμοί, ο Οργανισμός Φαρμάκων και η CDC, θα μετακινηθούν. Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αποφασίστηκε να μετακινηθεί στο Άμστερνταμ οργανισμός με βάση το άρθρο 50 της συνθήκης και με βάση τη διαδικασία που είχαν συμφωνήσει στις 22 Ιουνίου του 2017 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Αμέσως μετά η Κομισιόν που έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας έκανε μια νομοθετική πρόταση χρησιμοποιώντας τη συνήθη ε, νομοθετική διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία δεν ε, αναστέλει τα πράγματα περιτά και το Άμστερνταμ επιλέγει με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Μιλάμε ε, για εργαζόμενους ε, επιτόπου, ας πούμε, υψηλού επίπεδου. Το προτιμάει και ο αίμα. Και ε, υπάρχει και το σκύπολ, το αεροδρόμιο, το οποίο μπορεί να φέρει τις φαρμακευτικές εταιρείε και του τους εργαζόμενους τους πολύ κοντά στον οργανισμό φαρμάκων. Σε χρόνο τετέ. Όπως και για οργανισμού, οργανισμούς κινητικότητα ε, είναι ένα πρόβλημα. Από την πρώτη μέρα, και πρέπει να σας πω ότι εγώ ήρθα σε επαφή από την πρώτη μέρα με τον ε, Υπουργό μου, ε, αμέσως μετά τον Brexit έκανα λόμπι για να μετακινηθεί ο οργανισμό στο Άμστερνταμ, στις Καλοχώρε. Και δεν νομίζω ότι το να εμπλέξουμε το Κοινοβούλιο στην επιλογή των ε, οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σωστό. Το Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες και είναι συνομοθέτης. Δεν είμαστε μία επιλογή, μία εφορευτική επιτροπή, μία επιτροπή που επιλέγει γενικά μέλη ή επιλέγει πράγματα. Υπάρχουν επίσης ε, διαφορές. Ε, υπάρχουν μεγάλες και μεγάλες χώρες, χώρες με μεγάλο και μικρό πληθυσμό. Οι χώρες με μικρό πληθυσμό θα, ήταν, θα μειονεκτούσαν. Ε, μάλιστα αυτό συνέβη την περασμένη εβδομάδα σε μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ελπίζω μαζί να παίρνουμε τι σωστέ αποφάσει. Μιλάμε για δημόσια υγεία και την προστασία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να στραφώ επίση στον ε, συναδελφό μου στα δεξιά, στην Ολλανδία. Ε, με αυτόν τον τρόπο ανακτούμε την εμπιστοσύνη μα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Λίζα. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Λαβία για την εξαιρετική δουλειά που έκανε για το θέμα αυτό. Και θέλω ξεκάθαρα εδώ να, να υποστηρίξω αυτούς που λένε ότι αυτή η διαδικασία δεν προχωράει. Ο κλήρος επιλέγει ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά δεν έπρεπε καν να το έχουμε επιτάπητος, έπρεπε να είμαστε στη συναπόφαση, αλλά το, το Συμβούλιο αποφάσισε την κλήρωση. Και πρέπει να προσθέσω ότι η διαδικασία που έγινε πριν από την ε, όλη ψηφοφορία αυτή, ε, την ε, κλήρωση, ήταν πολύ αντιδημοκρατική. Δεκαετίες συζητούμε πώς θα δημιουργήσουμε, πώς θα χτίσουμε δημιουργία στην Ευρώπη. Και μετά υπάρχει ένα, μια συμβαστική πρόταση που λέει ότι αν ε, πρέπει να ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία στο Συμβούλιο, θα γίνει με ειδική πλειοψηφία. Και αυτό είναι σκόπιμο. Κάθε χώρα έχει μία ψήφο, αλλά για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση δεν χρειαζόμαστε μόνο την πλειοψηφία των χωρών, αλλά και την πλειοψηφία του πληθυσμού. Οπότε λαμβάνεται υπόψη το ότι έχουμε κράτη τα οποία εκπροσωπούνται και τα οποία έχουν δημοκρατία. Και με την πρόταση της Κομισιόν, η Κομισιόν δηλαδή έχει την πρώτη ευθύνη, είναι απαράδεκτο οι θεματοφύλακες της ε, δημοκρατίας να κάνουν τέτοιες προτάσεις και βάζουν αυτή την πρόταση στο τραπέζι. Το, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο έχουν τις ίδιες ψήφους με τη Γαλλία και την Ιταλία. Αυτά ε, ουσιαστικά καταρρύπτουν όλα όσα έχουμε αποφασίσει τόσα χρόνια. Αγαπητή Κομισιόν, αγαπητό Συμβούλιο, τα κάνατε μαντάρα. Και αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Και γι' αυτό εγώ πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να πω αν έχουμε συναπόφαση να δούμε πού είναι η πλειοψηφία και πού θέλει η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών να πάει ο οργανισμός. Εγώ θα υποστήριζα το, Στρασβούργο και λυπάμαι που η γαλλική κυβέρνηση ε, πήρε τόσο ανόητη θέση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βλέπω και την αναγκαιότητα να μην δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα. Πρέπει να έχουμε μια κανονική απρόσκοπτη μεταβατική περίοδο και πρέπει να δεχτούμε ότι τώρα ο οργανισμός θα είναι στο Άμστερνταμ και να φροντίσουμε ότι αυτό θα γίνει γρήγορα με όλα τα θέματα που ανέφερε και ο Τζοβάνι Λαβία στην εκθεσή του. Αλλά το λέω σαφώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει πριν εδώ να μας πούνε να μας εξηγήσουν και να μας δηλώσουν ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει καμία, για καμία είδους επιλογή η ίδια διαδικασία. Γιατί την ευθύνη θα την έχουν αυτοί μετά. Και νομίζω ότι θα πρέπει και στον κύριο Ζέμαερ και στον κύριο Γιούνκερ να το πούμε αυτό. Δεν γίνεται και δεν πρέπει να επαναληφθεί, γιατί αλλιώς θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Η κυρία Μποναφέ. Grazie, Presidente. Πρόεδρε, ως όργανο που εκπροσωπεί τους πολίτες και που λογοδοτεί στους πολίτες, εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά και συμφωνώ με την αμηχανία των συναδέλφων για τους τρόπους με τους οποίους επελέγει, επιλέγει νέα έδρα του οργανισμού φαρμάκων. Δηλαδή με λοταρία, με, ε, στην τύχη το αφήσαμε. Δηλαδή. Και όμως μιλάμε για έναν οργανισμό που έχει μεγάλη σημασία για την τύχη των πολιτών, αποφασίζει για την ασφάλεια των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε. Και επομένως ε, και εγώ συμφωνώ ότι ίσως αξίζει να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμό σε εμά. Η διαδικασία λοιπόν, συμφωνώ, είναι απαράδεκτη. Πρέπει να την συζητήσουμε και να εμβαθύνουμε σε αυτή. Έδειξε την αδυναμία λήψης απόφασης των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για σημαντικά θέματα για τη ζωή των πολιτών και έδωσε επιχειρήματα σε όλους όσους πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη. Επομένω, συμφωνούμε, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτέ τι ε, διαδικασίε, πρέπει να τι αμφισβητήσουμε εν το βάθη. Το όργανο το οποίο εκπροσωπεί του πολίτε, επειδή ακριβώ του εκπροσωπεί, θα πρέπει να εμπλακεί. Και δεν μπορεί να εμπλακεί ε, πάνω σε τετελεσμένα. Αυτό το προβλέπουν οι συνθήκε. Νομίζω λοιπόν ότι η διαθεσμική συμφωνία που αντίθετα δεν δίνει κανένα ρόλο στο κοινοβούλιο είναι μια συμφωνία λανθασμένη. Και να περάσω τώρα σε ένα άλλο σημείο το οποίο αξίζει προσοχή μα, Μιλήσαμε για μια προσωρινή μεταφορά, εν αναμονή τη μόνιμη μεταφορά τη Έδρα. Και εγώ θα ήθελα με περιέργεια να μάθω τι σημαίνει αυτό σε οικονομικού όρου για την, τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής και για να είμαστε σίγουροι και να είναι σίγουροι και αυτοί που δουλεύουν στον οργανισμό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το χρονοδιάγραμμα θα γίνει σεβαστό. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Θα έλεγα πριν την ψηφοφορία να σκεφτούμε να κάνουμε μια ακρόαση για αυτούς που κάνανε την αξιολόγηση των υποψηφιωτήτων, ούτω ώστε να δούμε ποια είναι τα κριτήρια και να είμαστε σε θέση αν μπορούν να, γίνουν, να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν σεβαστά. Ευχαριστώ. Και τώρα, η Κομισιόν, ε, ο κύριος Χένινγκ ε, από τη Γενική Γραμματεία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Χένινγκ Κλάους είναι το όνομά μου. Να σας πω το εξής τι να κάνουμε που το πλαίσιο για να αποφασίσουμε για την ε, έδρα ενός οργανισμού είναι κοινή προσέγγιση που υπογράφηκε, ε, συμφωνήθηκε από τα τρία θεσμικά όργανα το 2012. Δεν υπάρχει τίποτα το κενοφανές μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι η Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν έχει δυνατότητα να πάρει απόφαση για την έδρα των μελλον... τις μάλλον των δύο αυτών οργανισμών. Απλώς βοήθησε τα κράτη-μέλη στην διαδικασία. Το, και αυτό που έκανε το καλοκαίρι ήταν να αξιολογήσει τις 28 προσφορές από τα κράτη-μέλη και για τους ε, δύο οργανισμούς. Δεν ε, κατάρτισε ούτε συστάσεις ούτε shortlist υπέρ, ε, για τη μία ή την άλλη έδρα των δύο οργανισμών. Η Κομισιόν έκανε απλώ την αξιολόγηση. Υπέβαλε την αξιολόγησή τη στα κράτη-μέλη και συνεχεία τα κράτη-μέλη ήταν απόλυτα ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν ή να μην χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση τη Κομισιόν κατά τη λήψη τη απόφασή του. Για την διαφάνεια τώρα, να σα πω δύο λόγια. Νομίζω 31 Ιουλίου ήταν η καταληκτική ημερομηνία και όταν μπήκαν οι προσφορές από τα κράτη-μέλη, υπευλήθηκαν μάλλον, ε, ανέβηκαν και στην ε, ιστοσελίδα ε, από το Συμβούλιο. Και συνεχεία την ίδια μέρα έβαλε και τις προσφορές στην δική της ιστοσελίδα Κομισιόν. Να, τι έχω να πω για τη διαφάνεια. Και επίσης, για να απαντήσω στον εισηγητή, τον κύριο Λαβία, η κοινή προσέγγιση είναι μια πολιτική, νομικά μη δεσμευτική συμφωνία και όμως είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αποφασίζουμε τέτοια πράγματα. Η Κομισιόν είχε σκεφτεί ότι για λόγους ασφάλειας, νομικής ασφάλειας, ασφάλειας σχεδιασμού, αυτές οι δύο προτάσεις που έχετε ενώπιό σας έπρεπε να γίνουν. Καταρχάς, στον ιδιωτικό καονισμό ε, της ε, ΕΜΠΑ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, το Λονδίνο αναφέρεται στο κανονισμό. Υπήρχε λοιπόν ε, ανάγκη να κάνουμε μια τροποποιητική πρόταση και για λόγους συνέπειας και για να ξεκαθαρίσουμε νομικώς πώς ότι η ημερομηνία της μεταφοράς, δηλαδή όταν αρχίζει να ισχύει η νέα έδρα, είναι η 31η ε, Μαρτίου του 2019 το αργότερο. Αυτό μπήκε για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και στις δύο ιδρυτικές πράξεις. Αυτό κάνει η Κομισιόν, αυτά έκανε η Κομισιόν. Δεν μπορώ να σχολιάσω τη διαδικασία περαιτέρω. Πρέπει να σας πω ότι υποβλήθηκαν, επαναλαμβάνω, ότι υποβλήθηκαν 28 προσφορές και για τους δύο οργανισμούς. Πολλές χώρες λοιπόν. Μπορεί να θεωρηθεί αυτό επιτυχία της διαδικασίας και όχι αποτυχία όπως υπόθηκε. φαίνεται ότι δίνεται μεγάλη σημασία στις ε, ανάγκες και στα συμφέροντα το, του προσωπικού και των ε, μελών των οικογενειών τους. Τώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για να γίνει αυτή η μεταφορά απρόσκοπτα. Και εμάς μας ενδιαφέρουν τα συμφέροντά τους ε, και η ευημερία τους. Υποστηρίζουμε και τους οργανισμούς και το προσωπικό σε αυτή τη διαδικασία. Κοιτάμε τον εσωτερικό κανονισμό, την κατάσταση του με τα σχολεία, εσωτερικό οργανισμό ενώ των δύο οργανισμών. Έτσι. Ο εισηγητή ζήτησε πληροφορίε για κάποια θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση. Σας παραπέμπω σε αυτό στις διαδικασίες, τις λεγόμενες building procedures που λαμβάνουν χώρα παράλληλα με αυτήν εδώ τη διαδικασία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου γιατί εγώ δεν έχω τα τελευταία νούμερα. Ίσως ε, ο εκπρόσωπος του οργανισμού φαρμάκων να μπορεί να σε ενημερώσει καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι από την προσωρινή έδρα στην μόνιμη έδρα, όλο αυτό το κόστος που ε, επισύρει αυτή η μεταφορά, θα πληρωθεί από τις ε, κάτω χώρες. Και αυτό υπήρχε ήδη στην Ολλανδική προσφορά. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να σε εκπλήξει κάτι τέτοιο η Κομισιόν δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσει κάποιου άλλου, δηλαδή της Ολλανδικής κυβέρνησης, εν προκειμένου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε να υποστηρίξουμε την Ολλανδική κυβέρνηση και να ενημερώσουμε εσά για την ε, διαδικασία και τα περαιτέρω βήματά της και να παραμένουμε σε στενή επαφή. Ε, ήδη υποστηρίζουμε όσο μπορούμε τον Οργανισμό Φαρμάκων και την ΕΜΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, στο μεταξύ την ενδιάμεση δηλαδή φάση. Τώρα, ο κύριος Βότιον ε, από την ΕΜΑ, τον Οργανισμό Φαρμάκων. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μία εισαγωγική δήλωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το follow-up μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα και οι επιπλοκές στην έμα είναι ε, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μετά το 1996. Πρόκειται για ειδικέ συνθήκες και ε, εξωτερικές συνθήκες οι οποίες μας επιβάλλουν ένα ζήτημα που το οποίο πρέπει να χειριστούμε. Μετά από το δημοψήφισμα αρχίσαμε την προπαρασκευαστική μας εργασία και αυτό αυτό αφορά και την λήψη απόφασης για την έδρα στις 20 Νοεμβρίου και είχαμε συζητήσεις και με τις Ολλανδικές Αρχές για το προσωρινό κτίριο και το μόνιμο κτίριο στη συνέχεια. Θα ήθελα να τονίσω ότι ότι δεν σημαίνει ότι στις 29 Μαρτίου είμαστε στο Λονδίνο και 30 Μαρτίου θα βρισκόμαστε στο Άμστερνταμ. Χρειάζεται πολλής προγραμματισμός και συζητήσεις έτσι ώστε ε, χάρη των ασθενών της Ευρώπης θα προσπαθήσουμε να χειριστούμε το ζήτημα κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο τώρα ως προς τη διαδικασία την οποία ανέφερε το Κοινοβούλιο, η επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων προβλέπει διαδικασία προσωρινής έδρας τη στιγμή που δεν θα υπάρχει οριστικό κτίριο μέχρι τις 30 Μαρτίου του 19. Αυτό αφορούσε την Ολλανδία. Μετά την απόφαση για την ε, έδρα συζητήσαμε στην Ολλανδία με τους συναδέλφους, ε, είχαμε εναλλακτικέ ε, που είναι μέρος του διαγωνισμού στο παράρτημα που έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και θεωρήσαμε ότι αυτές οι επιλογές δεν μπορούσαν να εγγυηθούν τη συνέχεια των εργασιών της ΕΜΑ. Είχαμε και μια τρίτη προσφορά Τώρα έχουμε μία τέταρτη εναλλακτική που είναι η καλύτερη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων πιστεύει ότι μπορεί να δεχτεί αυτή την τέταρτη προσφορά γιατί δεν υπάρχει άλλη καλύτερη εναλλακτική που να καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού φαρμάκων και θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Αν κινηθούμε πέρα από τον Ιανουάριο του 2018, δεν θα Έχουμε έτοιμα γραφεία την 1η Ιανουαρίου του 19 στο προσωρινό κτίριο. Γιατί φυσικά θα πρέπει να εξοπλιστεί το ε, κτίριο και φυσικά να πληρούνται και οι προδιαγραφές ασφαλείας και ταυτοποίησης. Άρα θα έχουμε μία διπλή κίνηση. Όταν έχετε προσωρινό κτίριο είναι σαφές ότι θα έχετε καταρχήν τη μεταφορά της EMA στην προσωρινή έδρα και από την προσωρινή στη μόνιμη. Οι Ολλανδικές αρχές μας είπαν, και αυτό αναφέρεται στο παράρτημα του ε, Μνημονίου ότι θα καλύψουν πλήρως το κόστος για τη μεταφορά από, τη μεταφορά, από την προσωρινή έδρα στη μόνιμη λαμβάνοντας υπόψη και την εγκατάσταση την τελική έδρα. Άρα δεν θα δαπανηθούν χρήματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη μεταφορά από την προσωρινή στη μόνιμη έδρα. Όμως αυτή η διπλή κίνηση δημιουργεί περισσότερες προκλήσεις από αυτές που ήδη έχουμε. Θα πρέπει για είναι δοκιμές των οπτικοακουστικών μέσων και στα δύο κτίρια και στο προσωρινό και στο μόνιμο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα επιχειρηματικό σχέδιο συνέχειας, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα. Λαμβάνοντας υπόψη και την τέταρτη επιλογή που θα πρέπει να καταστεί λειτουργική. Αυτή η επιλογή προβλέπει το ίμιση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που έχουμε στο Λονδίνο. Θα έχουμε λιγότερα γραφεία δηλαδή και λιγότερους χώρους συνεδρίασης. Γι' αυτό θα προβάλλουμε αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο συνέχειας, δίνοντας προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες για την ε, επίβλεψη και εποπτεία καθώς και χρήση των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Οι Ολλανδικές αρχές μας υποσχέθηκαν ότι πέρα από από τους χώρους συνεδριάσεων στο προσωρινό κτίριο θα μας ε, παράσχουν και επιπλέον χώρο στα ξενοδοχεία που βρίσκονται κοντά. Και θα πρέπει να τηρήσουν αυτή την υπόσχεση. Ως προς την ημερομηνία τώρα και κατά πόσο θα τηρηθεί ή όχι. Εμείς χρειαζόμαστε ασφάλεια αυτό σημαίνει 30 Μαρτίου 19. Ο οργανισμός φαρμάκων θα πρέπει να προγραμματίσει να φύγει από το Λονδίνο στις 30 Μαρτίου το 19 το αργότερο. Εάν τώρα μετακινηθεί αυτή η ημερομηνία θα έχουμε δυσκολίες για να βρούμε χώρο γραφείων. Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις με τις Ολλανδικές Αρχές θα πρέπει να τηρήσουμε την ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2019 για την προσωρινή έδρα έτσι ώστε να είναι λειτουργική η προσωρινή έδρα μέχρι αυτή την ημερομηνία για να μπορέσει να μεταφερθεί η EMA μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2019 έτσι ώστε να γίνει τελική μεταφορά στις 30 Μαρτίου του 2019. Εάν αρχίσουμε να αλλάζουμε τις ημερομηνίες τότε δημιουργούμε δυσκολίες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για να λειτουργήσει, αλλά και για το προσωπικό που πρέπει να γράψει τα παιδιά του στο σχολείο, που αγοράζει σπίτια ή πουλάει και ε, ψάχνει εργασία και για τα μέλη της οικογένειας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μετακινήσουμε, να μετακινήσουμε την ημερομηνία της 30ης Μαρτίου 19. Επίσης, έγινε λόγος για την έδρα ε, η έδρα, η συμφωνία περί έδρας ε, θα υπογραφεί το συντομότερο δυνατόν. Και θα δώσουμε τελική μορφή στις συζητήσεις το αργότερο τα τέλη Μαρτίου του 2018, έτσι ώστε να αρχίσει η διαδικασία συνεννόησης με την Ολλανδική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι θα υπογράψουμε μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2018. Αυτό που έχει σημασία βεβαίως πέρα από το χρονισμό είναι και το περιεχόμενο. Γιατί με αυτή την κατάσταση καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνεται το έργο μας. Δηλαδή δεν μιλάμε για μία εξ αρχή σύσταση οργανισμού. Γι' αυτό θεωρούμε ότι οι Ολλανδικές Αρχές θα πρέπει να μας δώσουν την καλύτερη δυνατή ε, δυνατότητα συνέχειας, κυρίως για το προσωπικό. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λαβία για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξη και για την ταύτιση απόψεων. Θέλω να επανέλθω στην τη συζήτηση σε κάποια στοιχεία που σχετίζονται περισσότερο με τις διευκρινήσεις που μας έδωσε η και ο εκπρόσωπος της ΕΜΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Καταρχάς το πρώτο. Αυτή η κοινή δήλωση δεν αναφέρθηκε στην πρόταση της Κομισιόν. Και δεν την ήξεραν αυτή η κοινή δήλωση οι περισσότεροι βουλευτέ. Σήμερα τη μάθανα. Και παρόλα αυτά καθόρισε όλη τη διαδικασία. Σίγουρα με την κοινή δήλωση εκχωρήθηκε η αρμοδιότητα στο Συμβούλιο, αλλά δεν δόθηκαν καθόλου λεπτομέρειες για την διαδικασία. Καθόλου λεπτομέρειες σε, αυτή την, σε αυτό το joint statement. Και αυτό το joint statement, μάλλον αυτή η διαδικασία, δεν είναι σύμμορφη με το βάρος, το ειδικό βάρος των χωρών. Και τελικά η επιλογή ήταν μια μη επιλογή, μια και τελικά έγινε κλήρωση για να αποφασίσουμε τελική έδρα. Είναι ξεκάθαρο και μου κάνει εντύπωση που η Κομισιόν δεν μας ενημερώνει καθόλου για το πώς προχωρούν οι εργασίες για την προσωρινή έδρα, αλλά ούτε και για την μόνιμη έδρα. Γιατί αντικειμενικά αυτό θα καθορίσει όλη τη διαδικασία. Φυσικά καταλαβαίνω ότι η Ολλανδική κυβέρνηση θα κάνει τις εργασίες και θα ε, φροντίσει τόσο ώστε οι δεσμεύσεις να γίνουν σεβαστές. Αλλά θα πρέπει οι δεσμεύσεις αυτές να τις παρακολουθεί κάποιος. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βρεθεί στη θέση και δεν να πρέπει να δικαιολογήσει γιατί δεν πήγαν καλά τα πράγματα και γιατί δεν μπορούν να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για τον οργανισμό. Επίσης, ό,τι αφορά τις προθεσμίες, τα χρονοδιαγράμματα, προκύπτει ξεκάθαρα από την τοποθέτηση του προσώπου της ΕΜΑ ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σκεφτεί κανεί ότι στι 29 θα είναι όλοι στο Λονδίνο και στι 30 θα, μεταφερθούν, θα διακτενιστούν στην νέα έδρα. Από την άλλη όμω, για να λειτουργεί η αίμα, δεν θα πρέπει να αλλάξει η ημερομηνία αυτή. Επίσης, στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου θα πρέπει να προβληματιστούμε για αυτή την κοινή δήλωση, για αυτό το joint, joint statement. Γιατί εγώ δεν πιστεύω και με επιβεβαίωσαν και οι συναδελφοί μου ότι αποφάσεις τέτοιου βελληνικού. που δεν είναι τεχνικές αποφάσεις, αλλά που είναι υψίστως ε, πολιτικές, δεν πιστεύω ότι τέτοιε αποφάσει θα πρέπει να γίνονται χωρί ε, χωρίς την εμπλοκή των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών λαών. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ, και είναι απόλυτη πεποίθησή μου, ότι μία ε, επιπλέον δήλωση του Κοινοβουλίου με βάση αυτό που θα ψηφίσουμε στην ε, Επιτροπή είναι σημαντική για να πάρουμε θέση στο θέμα. Και καλό όλου του και όλου για να συνεργαστούν και να συντάξουν από κοινού αυτή την πρόσθετη δήλωση. Δεν θέλω να είναι δική μου δήλωση, θέλω να είναι μία ε, δήλωση του Κοινοβουλίου, κοινή θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι 31 Ιανουαρίου, 11 το πρωί. Πάμε στο επόμενο σημείο. Η επιφυλακτικότητα και η μείωση της κάλυψης ε, των εμβολιασμών στην Ευρώπη. Η κυρία Σόμαρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλήξαμε σε ένα πολύ καλό κείμενο για το ψήφισμα, το οποίο καταγράφει όλα τα βασικά προβλήματα και την επιφυλακτικότητα και τη μείωση κυρίως των ε, εμβολιασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους από τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί πραγματικά η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική. Σίγουρα όλοι θα έχετε την ίδια ανησυχία για την επιφυλακτικότητα που υπάρχει απέναντι στους εμβολιασμούς, η οποία πρέπει να σταματήσει. Και η μείωση επίσης φαίνεται να υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Είναι μια ανησυχητική ιδιαίτερο εξέλιξη, γιατί όλο και μεγαλύτερο αριθμός ε, πολιτών αρνείται να εμβολιαστεί. Και βεβαίω αυτό είναι ο μόνο και ίσω από του καλύτερου τρόπου ε, πρόληψη ε, ασθενειών που έχουμε στην διάθεσή μα. Ε, τα εμβολιαστικά προγράμματα έχουν οδηγήσει από τι αρχέ του 20ου αιώνα στην μείωση σημαντικών πανδημιών σε περιοχές του κόσμου, της Ευρώπης ε, κατα, ε, εξαφανίστηκε ουσιαστικά η πολιομιλίτιδα ε, από το 80 έχουμε πραγματικά πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οι εμβολιασμοί μπορεί να θεωρούνται ότι δεν είναι απαραίτητοι πλέον, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να παραμείνουν μη απαραίτητοι. Εκτός αν οι πολίτες παραμείνουν τόσο δυστακτικοί, γιατί θα αρχίσουν να υπάρχουν ε, ξανά ε, ασθένειες τις οποίες ε, ήδη εδώ και πολλά χρόνια έχουμε καταφέρει να απαλείψουμε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε, έχουμε εξαφανίσει ουσιαστικά κρούσματα ασθενειών. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, σας διακόπτω. Παρακαλώ, λίγη ησυχία στην αίθουσα μπορούμε να έχουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. πραγματικά οι διάφορες ασθένειες, ας πούμε, η ερυθρά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους ε, πολίτες και ακριβώς λόγω των εμβολιασμών τους έχουμε, έχουμε καταφέρει να ε, απαλείψουμε τέτοιου είδους ασθένειες και νομίζω ότι είναι πραγματικά ανεύθυνο όταν οι γονείς δεν κάνουν εμβόλια στα παιδιά τους επειδή θεωρούν ότι ε, εντάξει αφού όλα τα υπόλοιπα είναι εμβολιασμένα δεν χρειάζεται να εμβολιαστεί το δικό μου και υπάρχει και αυτή η φήμη που λέει ότι ε, τα εμβόλια προκαλούν άλλες ασθένειες. Τα εμβόλια δεν διακυβεύουν την υγεία των παιδιών, δεν είναι περιτά και δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των, της φαρμακοβιομηχανίας, είναι προς το συμφέρον όλων μας. Και ακριβώς επειδή, ε, αν δούμε μάλλον την, κατάσταση τώρα, ακριβώς επειδή υπάρχει και τεράστια μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από κάθε είδους χώρα, που δεν ξέρουμε αν υπάρχει σταθερός εμβολιασμό ή οποιοδήποτε είδου εμβολιασμό, καλό θα ήταν βλέποντας την κατάσταση να είναι σαφέ σε όλου μα ότι πρέπει να φροντίσουμε οι πολίτες να αρχίσουν και πάλι τακτικά να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, εξτρατείες ενημέρωσης, όπως ζητά και η Κομισιόν από το Συμβούλιο των Υπουργών, είναι πραγματικά τεράστια η ευθύνη των κυβερνήσεών μας. Ίσως να αποκοιμηθήκαμε λίγο και να το ξεχάσαμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και επίσης, ευρωπαϊκά θα πρέπει ίσως υποχρεωτικά να επιβάλλουμε κάποιους εμβολιασμού. Στην ε, Γερμανία για τις βασικές ασθένειες ο εμβολιασμό είναι υποχρεωτικός. Κάθε χρόνο μιλούμε για την αντιμικροβιακή αντίσταση και περίπου 25.000 ετησίω στην Ευρώπη πεθαίνουν από ασθένειες που θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει. Γι' αυτό ο εμβολιασμό θα μπορούσε όντω να αποτελέσει ελπίδα πάληψη τέτοιων φαινομένων. Οπότε ζητούμε από τα κράτη-μέλη και από την ε, Κομισιόν να συνεργαστούν και πολύ γρήγορα να εκπονήσουν ένα σχέδιο δράση, γιατί πραγματικά θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Thank you. Now, uh, Mrs. Εγώ ευχαριστώ. μάλλον. Ε, κυρία Τζεντήλε, ε, η ιστορία μας δίνει εντυπωσιακά νούμερα. Η χρήση των εμβολίων στο παρελθόν μας επέτρεψε να εξαλείψουμε σοβαρότερες ασθένειες. με σοβαρότες επιτυχίες σε ό,τι αφορά το κέρδος ανθρώπινων ζώων. Η πρόσφατη ιστορία όμως, αντίθετα, μας δίνει κάποια άλλα δεδομένα εξίσου σημαντικά που αντισταθμίζουν αυτά που σας έδωσα πριν για το παρελθόν. Το 2017 ε, έγινε μια... Είχαμε μια νέα επιδημία πολυ... πολυομιλίτιδας στην Ευρώπη. Στη χώρα μου 450 άτομα μολύνθηκαν από τον ιό. Είχαμε κάποιους θανάτους, και ένα ποσοστό ανθρώπων αρρώστησε στις, στα πρώτα στάδια της ζωής του. Αυτό τι μας δείχνει. Ότι είμαστε εκτεθειμένοι ε, σε μία πιθανότητα άλλων επιδημιών. Άρα θα πρέπει να εγγύψουμε με προσοχή στο θέμα αυτό. Και ελπίζω να συμφωνήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά και ελπίζω σε όλο το Κοινοβούλιο, ότι υπάρχει ανάγκη να θέσουμε αυτό το ερώτημα. Σε ευρύτατο επίπεδο. Κυρίως για να υπευθυνοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την Κομισιόν για να ξεκινήσει ένα τεράστιο ενημερωτικό πρόγραμμα και πρόγραμμα κατάρτισης παράλληλα σε όλα τα κράτη-μέλη, κυρίως τα κράτη-μέλη που είναι τα πιο τροτά, τα πιο που είναι ανοιχτά, αν θέλετε, σε fake news, σε ψεύτικες πληροφορίες, ε, σε ειδήσει χωρίς κανένα επιστημονικό, ας πούμε, υπόβαθρο. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ας το δούμε με την ευαισθησία του καθένας. Και ας αναρωτηθούμε και εμείς, αλλά και ας ρωτήσουμε την Κομισιόν, όχι μόνο να υπάρξει μια πολύ μεγάλη δέσμευση, γενναιόδορη δέσμευση, γιατί θα πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα επίγνωση, θα πρέπει να υπάρξει μια νέα αφύπνιση και υπάρχει ανάγκη να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο την έρευνα, για να υπάρξουν νέα εμβόλια, για να εξαλείψουμε αρρώστιες επίσης ε, σημαντικές. Παραδείγματο χάρη τον, ε, τον ιό ο οποίος πλήττει τον, ε, τη μήτρα των γυναικών και τον, τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων. και θα πρέπει να βρεθούν και συστήματα αγοράς του εμβολίου, ούτω ώστε να μειωθεί το κόστος που θα πρέπει να καταβάλει το, κάθε κράτος μέλος για την αγορά των εμβολίων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την υγεία των παιδιών και κυρίως των κοριτσιών μας, ε, που είναι το πιο σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Σε μια Ευρώπη των πολιτών, δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτό το τόσο μεγάλο θέμα και να αγνοούμε αυτό το τεράστιο δράμα που έλαβε χώρα την περασμένη χρονιά. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ υποστηρίζω την ε, έκθεση αυτή. Μιλούμε για τους ε, ε, εμβολιασμού στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και έχω την εντύπωση ότι οι εμβολιασμοί από τον 19ο αιώνα έχουν εφευρεθεί. Ήταν πάρα πολύ δημοφιλής τον 20ο αιώνα και οι εμβολιασμοί αυτοί μας έχουν ε, βοηθήσει να εξαλείψουμε ασθένειες όπως η ε, πολιομιελίτιδα η Ερυθρά. Ε, αλλά τώρα υπάρχουν νέε πηγές αυτών των, αυτών των ασθενειών. Για ασθένειε, μάλιστα τι έχουμε ξεχάσει εδώ και κάποια χρόνια, ακριβώ λόγω των πολύ δημοφιλών εμβολιασμών. Στο σχέδιο έκθεσης δείχνουμε ότι τα δεδομένα αυτά από τα κράτη-μέλη μας δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά κενά σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμού. Οι εμβολιασμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Είναι απαραίτητοι να, για να εγγυηθούμε την υγεία των πολιτών. Και πραγματικά χρειάζεται όντως ένα ευρύ σχέδιο δράσης ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την επιφυλακτικότητα που δείχνουν οι πολίτες στους εμβολιασμούς. Γιατί όμως προκύπτουν αυτή η δισταγμή απέναντι στα εμβόλια. Κυρίως γιατί οι πολίτες λαμβάνουν λανθασμένες πληροφορίες για τα εμβόλια. Φαίνονται σαν να είναι επιστημονικές οι πληροφορίες αυτές, αλλά δεν είναι και πραγματικά θα πρέπει να εναρμονίσουμε τα σχέδια δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την επιφυλακτικότητα που δείχνουν οι πολίτες απέναντι στα εμβόλια. Ευχαριστώ. Η κυρία Μιούλερ εκ μέρους της κυρίας Μάισνερ. Ε, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους τη κυρίας Μάισνερ, είναι δυστυχώς ε, άρρωστη. Βεβαίως υποστηρίζουμε πλήρως την έκθεση αυτή και εμείς θεωρούμε ότι ο, ο βαθμός μειώνεται στην Ευρώπη και είναι πολύ ανησυχητικό. Ε, ε, μπορεί να θεωρείται βέβαια όχι καθημερινό ίσως πρόβλημα, αλλά για την, ίσως να πρέπει όντως να ενταχθεί ένας ε, υποχρεωτικός εμβολιασμό στην επικράτεια της Ευρώπης. Θα πρέπει βέβαια να δούμε και το κόστος για τα συστήματα υγείας Ας πούμε, οι παιδικές ασθένειες ε, αυξάνονται συνέχεια, η ανεμοβλογιά, η λαρά, η ερυθρά, είναι πραγματικά μεγάλο ε, βάρος αυτό και για, την, για τα συστήματα υγείας από πλευράς κόστους και για την υγεία των ε, πολιτών. Είδαμε τι έγινε στην Ιταλία πέρσι. Εγώ είμαι πολύ περήφανη που και τα δύο μου εγγόνια είναι εμβολιασμένα και που οι γονείς τους ε, δεν παρακολουθούν, δεν ακολουθούν μάλλον αυτή την εκστρατεία που είναι κατά των εμβολιασμών και υποστηρίζουμε απολύτως την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Uh, uh, Πρόεδρε, συμφωνώ με εκείνους που ήδη μίλησαν για αυτό το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε. Αλλά με ανατακτά διαστήματα το συζητάμε όταν ξεσπάει οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ασθένεια, μια ασθένεια που πιστεύαμε ότι είχε εξαλειφθεί στην Ιταλία, στη Ρουμανία και στη Γερμανία, μέχρι το Φεβρουάριο του 2017 υπήρχαν 1.500 ε, νέες περιπτώσεις ηλαράς και το 75% από αυτές ε, οφείλεται σε έλλειψη εμβολιασμού. Η εμβολιαστική κάλυψη πέφτει, το ποσοστό πέφτει και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί λόγω του υπερβαλλικού κινδύνου που συνδέεται με τον εμβολιασμό, υποτίθεται, και λόγω του κινδύνου των μεταδοτικών ασθενειών δεν μπορούμε να περιμένουμε να πεθάνουν 200 άτομα λόγω ηλαράς πριν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να πούμε τα, πράγματα, τα πράγματα με το όνομά του, τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αυτέ οι παραπλανητικέ πληροφορίε, αυτά τα ψέματα, μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Και εγώ είμαι μητέρα και ξέρω πολύ καλά ότι θα πρέπει να έχουμε καθαρά εμβόλια καθαρά προγράμματα εμβολίων που δίνουν και ευελιξία στους γονείς. Αλλά μέχρι εκεί θα πρέπει να ανασκευάσουμε όλους αυτούς τους γελίους μύθους για το τι υποτίθεται προκαλούν ε, τα εμβόλια. Οι παρενέργειες είναι πολύ σπάνιες από τα εμβόλια. Και δεν έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική ακόμα για να καταπολεμήσουμε την υπατήτασή, ε, την φυματίωση ε, και τον ιό του AIDS. Γι' αυτό κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, κάνει, να ξεκινήσουν, και στα κράτη-μέλη μαζί βέβαια, να ξεκινήσουν μια μαζική ενημερωτική εκστρατεία και ένα σχέδιο δράση για να καταπολεμήσουν τη μείωση του εμβολιασμού. Όσο τα κράτη-μέλη και οι υπουργοί αγνοούν τα δεδομένα και ακούν τις ΜΚΟ και ορισμένους ας πούμε θειασότες οι οποίοι καταπολεμούν τα εμβόλια εξ επαγγέλματος δεν θα αλλάξει τίποτα το μπαλάκι είναι στα χέρια των κρατών μελών, ειδικά των κρατών μελών. Η Κομισιόν φυσικά έχει αρμοδιότητε, αλλά θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στην πόρτα μα. Ο επόμενο ομιλητή εκπροσωπεί. Η επόμενη ομιλήτρια εκπροσωπεί τον κύριο Λαφρο, ε, Λαφρόντε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εκπροσωπώ τον κύριο Λα... Αφρόντε. Συμφωνώ με πολλά που ακούσαμε. Υπάρχουν και όμως και πράγματα που με βρίσκουν αντίθετη. Το, φάρμακο, το εμβόλιο για τη δευτερήτη, δακοκίτη, λαρά και ερυθρά ε, είναι πολύ σημαντικό. Και το εμβόλιο για την πολιομελίτιδα επίσης, αλλά μην γενικεύουμε. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί υπάρχουν και δισταγμοί και δυσπιστία. Γιατί έχουμε και τα fake news. Έχουμε φυσικά εμβολιαστικέ εκστρατείε που είναι παντελώ γελίε. Φερρυπίν εμβολιάσαμε τα άτομα, παιδιά ας πούμε, εναντίον της ε, πανόλης των χείρων. Και τελικά συνειδητοποίησαμε ότι το εμβόλιο αυτό δεν είναι πιο αποτελεσματικό από την παρακεταμόλη ας πούμε. Ας δούμε και τα νούμερα. Τα νούμερα είναι σαφή στη Δανία. Έχουμε 5 εκατομμύρια κόσμο και υπάρχουν 100 άτομα που πεθαίνουν κάθε χρόνο από έλλειψη εμβολιασμού, ενώ υπάρχουν 5.000 θάνατοι λόγω καπνού, λόγω καπνίσματος. Υπάρχουν επίσης και οι ηλικιωμένοι. Εάν εμβολιάσουμε τα παιδιά από 0 έως 13 ε, χρονών, ίσως θα σώσουμε 8 άτομα, ας πούμε, το οποίο είναι, τάξη. λίγα. Επίση πρέπει να δούμε τι γίνεται με του εμβολιασμού πιο ηλικιωμένων ανθρώπων. Υπάρχουν προβλήματα από τον εμβολιασμό. Είναι σαφέ ότι υπάρχουν προβλήματα. υπάρχει όμω βέβαια πρόβλημα και με τα fake news και με τα μέσα κοινωνική δικτύωση, ε, που διαδίδουν ας ψευδείς ειδήσει. Δεν το αρνούμε αυτό. Αυτό καταρρύπτει και υποσκάπτει την εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο εμβόλιο κατά τη φυματίωση, κατά τη ερυθρά κτλ. Θα πρέπει επίσης να είμαστε αντίθετοι στις ε, παραπλαντικές ε, ενημερώσεις. Παραδείγματο χάρη για τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων, κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι σαφέ. Αλλά δεν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται μια γενικευμένη εκστρατεία εμβολιασμού. Χρειάζεται πρόληψη και μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ε, εμβολίων. Ε, μεγαλύτερη διαφάνεια τη ζητούμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για το θέμα αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και των δημοσίων φορέων που υποσκάπτει την εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Αλλά συμφωνώ με την ουσία της έκθεσης. Πρέπει να υποστηρίξουμε ότι ορισμένα εμβόλια είναι εκ των όνου Αλλά δεν χρειάζεται να εμβολιαζόμαστε αντίον για να καταπολεμούμε όλες τις ασθένειες. Αυτό δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντορνάνο. Θέλω να συμφωνήσω κι εγώ. Γιατί στην Ευρώπη επανέρχονται κάποιες αρρώστιες ε, και εδώ παράλληλα βλέπουμε μία απροθυμία όλο και μεγαλύτερη απέναντι στον εμβολιασμό. Ε, προφανώς παρούσα και στη Γαλλία, τη χώρα μου. Ε, κάποια στοιχεία στο κείμενο είναι σημαντικά. Καταρχά, πρέπει να σεβαστούμε την, ε, το διαχωρισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Ε, Παράγραφο 7. Σημασία για να έχουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στα φάρμακα είναι να υπάρχει διαφάνεια. Στην παράγραφο 12 επίση, που καταγγέλουμε την ε, παραπληροφόρηση μέσω τη ε, κυκλοφορία πληροφοριών τύπου fake news, ε, ψευδών ειδήσεων. Επίση, πρέπει να ανησυχήσουμε για τι υψηλέ τιμέ κάποιων εμβολίων που παρόλα αυτά μπορούν να σώσουν ζωέ. Σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών εμβολιασμού σε μετανάστε και πρόσφυγε που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να, ξε, να ξεκαθαρίσω τη θέση μου και να την καταλάβετε. Φυσικά θα πρέπει να εμβολιάζουμε μαζικά, ούτως ώστε να εξαλείψουμε διάφορε ασθένειε και να αποφύγουμε επιδημίε που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πάρα πολλού θανάτου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όταν ξέρουμε ότι η Ερυθρά συνεχίζει να προκαλεί θανάτους. Παρ' όλα αυτά, μια και με ενδιαφέρει η κυριαρχία τη χώρα μου, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η προστασία και η βελτίωση τη ανθρώπινη υγεία εντάσσεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων ε, με βάση το άρθρο 6 της ε, Συμφωνία τη συνθήκη, μάλλον για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι υπάρχουν καλέ προθέσει εδώ, η Κομισιόν απλώ μπορεί να συμπληρώσει τι δράσει των κρατών μελών, να βοηθήσει, να υποστηρίξει. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό η νομικά δεσμευτικές ε, πράξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να ζητήσουν να υπάρξει νομοθετική εναρμόνιση και κανονιστική εναρμόνιση τη χώρα Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παράγραφο 19 αποκαλεί την Κομισιόν να προωθήσει την εναρμόνιση των χρονοδιαγραμμάτων για τον εμβολιασμό στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα. Επίση, θα καταθέσω τροπολογίε σε αυτό το κείμενο και θα ευχαριστήσω του ε, συντάκτε για τη βοήθειά του, και τα σχόλιά τους και τη συνεισφορά του εν πάση περιπτώσει. Κύριος Γραμματικάκης. Είναι πράγματι γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί ένα ιδιόμορφο κίνημα εναντίον των εμβολιασμών που έχει ευρωπαϊκές διαστάσει. Και βέβαια αυτό το κίνημα σχετίζεται με το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων, των fake news και συνεπώς είναι περίπλοκο και δύσκολο να το ελέγξει κανείς αφού έχει και πολιτικές ευαισθησίες. Υπάρχει όμως μια βεβαιότητα ότι τα κράτη-μέλη ελάχιστα μπορούν να πετύχουν από μόνα τους. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε σε δράσεις ευρωπαϊκού επίπεδου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στείλει κατά τη γνώμη μου ένα σαφές μήνυμα για τους κινδύνους του μη εμβολιασμού. Διότι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη ή ότι δεν φτάσαμε ποτέ στο φεγγάρι δεν βλάπτουν κανένα άλλο. Εκείνοι όμως που διαδίδουν τέρατα και σημεία εναντίον των εμβολιασμών βλάπτουν το διπλανό τους. Θέλω να πω δύο κουβέντες και να τελειώσω για τον εμβολιασμό κατά της Ιλαράς, που είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος με τα στοιχεία που έχω έχουν παρατηρηθεί 20.000 κρούσματα το 2017 σε όλη την Ευρώπη. 20.000 το υπογραμμίζω. Η Ελλάδα είχε 1.000 κρούσματα, η πατρίδα μου, ενώ δύο από αυτά ήρθαν θανατηφόρα. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι πραγματικός και ενδέχεται να διονγκωθεί. Αυτό θέλω να υπογραμμίσω αν δεν υπάρξει κατάλληλη αντίδραση. Ίσως πρέπει να δώσουμε εντολή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης νοσημάτων αναπτύξει μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική υπέρ του εμβολιασμού που υπήρξε μια μέγιστη επιστημονική πρόοδος των καιρών μας. Επίσης πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ψευδείς ειδήσει, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να δημιουργηθούν ευρωπαϊκά προγράμματα που να στοχεύουν στον εμβολιασμό κοινωνικών ομάδων που είναι πιο ευάλωτες ή παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού επικουρικά βέβαια πάντα στα εθνικά συστήματα υγείας. Το πρόβλημα μπορεί να μην μπορεί να εξαλειφθεί όλο, αλλά μπορεί να περιοριστεί σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω από ένα ανησυχητικό δεδομένο που ακούστηκε. Εμείς βλέπουμε στην Ευρώπη ότι πέφτει η εμβολιακή κάλυψη και ε, επανεμφανίζονται σοβαρότερες αρρώστιες που θεωρούσαμε ότι είχαν οριστικά εξαλειφθεί. Γιατί δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Σήμερα στην Ευρώπη πεθαίνουμε πάλι λόγω ηλαράς. Ευχαριστώ λοιπόν τους συναδέλφους που, που υπέβαλαν αυτό το ψήφισμα. Με βρίσκει σύμφωνη. Πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης. Και για να διευκολύνουμε ένα πρόγραμμα ε, ευρωπαϊκού εμβολιασμού, πιο εναρμονισμένου, αλλά και να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό πρόβλημα απροθυμίας για εμβολιασμό. Είναι ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα, ένα πραγματικό πρόβλημα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και να καταδικάσουμε την διάδοση ψεύτικων ειδήσεων, ε, παραπλανητικών και αντιεπιστημονικών για τον ε, εμβολιασμό, που επιβαρύνεται από, την, ε, από το γεγονός ότι ορισμένοι κάνουν εξαρτία κάτω του εμβολιασμού παίρνοντας πολιτική θέση, ας πούμε, πολιτική. Ορισμένοι φοβούνται ότι αν εμβολιάσουν τα παιδιά τους θα υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών. Ε, πείθονται από αυτές τις παραπλανητικές εκστρατείες. Ε, βεβαίως υπάρχουν μερικές φορές κάποιες αλήθειες, αλλά ορισμένοι είναι απόλυτα πεπισμένοι ότι όταν εμβολιαστεί ε, ένα παιδί θα έχει επιπτώσει αρνητικέ αυτό στη δική του υγεία, αλλά στην πραγματικότητα το να μην εμβολιαστεί έχει επιπτώσει στη δημόσια υγεία και στην υγεία των πιο ασθενών ανθρώπων. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σίγουρο το ότι ο εμβολιασμό σώζει ζωές και είναι ένα από τα πιο ε, σοβαρά μέτρα υγείας τα οποία θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη. Όμως δυστυχώς από μία πρόσφατη έρευνα φαίνεται στη Γαλλία ότι το 41% δεν συμφωνεί ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. το σύνολο αυτών που απάντησαν σε όλες τις χώρες αφορά 30%. Αυτό σημαίνει μείωση του εμβολιασμού, κάτι το οποίο έχει ολέθριες συνέπειες. Αν δείτε την έκθεση του Ιανουαρίου του 2018, βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει πολλά κρούσματα ηλαράς, κάτι το οποίο ε, οδήγησε σε 49 θανάτους μόνο σε ένα χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει γιατί ο εμβολιασμός είναι αναπόσπαστο μέρος μιας πολύ καλής ε, πολιτικής υγείας και στην ε, Φλάνδρα το αντιμετωπίζουμε αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα σε σχέση με τον εμβολιασμό. Όμως ε, οι γονείς είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν σωστές πληροφορίες και να συνειδητοποιούμε τους κινδύνους. Γι' αυτό υποστηρίζω αυτό το ψήφισμα πλήρως. Ο κύριος Πράτς. Ε, από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ, Γενικός Διευθυντής. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί το Κοινοβούλιο έδωσε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αντιδράσει σε σχέση με αυτό το ψήφισμα, το προσχέδιο. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό το ψήφισμα σε σχέση με τον εμβολιασμό. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τις κυρία Σόμερς Τζεντήλε και τους άλλους ε, συντάκτες. Ε, ήδη βλέπουμε ε, ότι υπάρχουν ίχνη ευλογιάς, ευλογιάς σε μία μούμια η οποία, ε, η οποία ανακαλύφθηκε και είναι 6.000 ετών. Αυτό είναι η καλύτερη δυνατή απόδειξη ότι θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση σε σχέση με τον εμβολιασμό των ανθρώπων. Και αυτό ιδιαίτερα στην Ευρώπη, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα σε σχέση με τον εμβολιασμό. Μόνο δύο κράτη-μέλη έχουν πλήρη κάλυψη εμβολιασμού σε σχέση με όλα τα εμβόλια όπως τα ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι προσυπογράφω αυτή την πρόταση και θεωρώ ότι η επιφυλακτικότητα ε, του εμβολιασμού, καθώς και η κάλυψη εμβολιασμού ε, αναφέρθηκε ήδη από τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Και γι' αυτό η Επιτροπή ε, υπέβαλε μία πρωτοβουλία μετά από ευρύ διαβούλευση και σε σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που λύγει μέχρι τις 15 Μαρτίου και Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη το νοσηλευτικό προσωπικό της Ενώσης Φαρμακείων Νοσηλευτών και γενικότερα νοσηλευτικού προσωπικού έτσι ώστε μέχρι ισότου υποβάλουμε την πρωτοβουλία να έχουμε καλύψει όλο αυτό το φάσμα διαβούλευσης. Επίσης, πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία θα είναι συνεχής. Ο εμβολιασμός έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπουμε πολλά κρούσματα και θα πρέπει φυσικά τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν πολύ καλά πώς θα πρέπει να επιβάλλουν ένα σχέδιο εμβολιασμού μέσα στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων υγείας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα ήταν μεγάλο σφάλμα να να θεωρήσουμε ότι η επιφυλακτικότητα εμβολιασμού είναι ένα θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να γίνει κοινή προσπάθεια από όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει πλήρης δέσμευση από την Επιτροπή να δώσει προστιθέμενη αξία σε αυτή την πρωτοβουλία και τον Απρίλιο φέτος θα προτείνουμε μία σύσταση του Συμβουλίου με την υποστήριξη μίας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε αυτή την ευρεία πρωτοβουλία όπως είπε και η κυρία Τορνανό καθώς και η κυρία Ζόμερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Uh, ευχαριστώ να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή. Η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι 30 Ιανουαρίου, 11 το πρωί. Επόμενο σημείο. Έκθεση προς ε, ε, έναν ανταγωνιστικό και βιώσιμο τομέα υδατοκαλλιέργειας. Να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Γκάμπους. Ευχαριστώ. Σήμερα σας παρουσιάζω την έκθεση γνωμοδότηση στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο βασικές ε, προκλήσεις, ε, την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος καθώς και τα ευεργετήματα από την αλληλεία και κατανάλωση αλλιευτικών προϊόντων στην ε, καθημερινή μας διατροφή. Όπως γνωρίζετε, με το πέρασμα του χρόνου υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση αλλιευμάτων και το σύνολο αφορά εισαγωγές 60% από άλλες χώρες, ενώ η δική μας υδατοκαλλιέργεια μας δίνει ένα 10% αλλιευτικών πόρων, γι' αυτό έχουμε πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Γιατί Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ευρεία κατανάλωση όλων των αλλιευμάτων και αυτό αφορά και την ποιότητα και την βιωσιμότητα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να συμμεριστούμε την εμπειρία μας με τις γειτονικές χώρες έτσι ώστε να βελτιώσουν τις πρακτικές τους για να γίνουν πιο βιώσιμες. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους αλληλείς, τους μεταποιητές, τους υδατοκαλλιεργητές έτσι ώστε να μπορέσουν να τηρήσουν αυτό το πλαίσιο της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και παράλληλα πώς μπορούμε να εξηγήσουμε στους καταναλωτές ότι η διατροφή με προϊόντα αλίας βοηθάει στην βιωσιμότητα του τομέα και αυτό αφορά τις δικές μας αλλιευτικές κοινότητες και την επιβίωσή τους. Θα πρέπει λοιπόν να προβάλλουμε μια πολύ καλή ποιότητα σε σχέση με τις κοινωνικές χώρες και αυτό αφορά και την ε, ευζοία μας και την ευζοία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις ε, χώρες ε, προέλευσης και όταν υπάρχει απόψυξη αλλιευμάτων θα πρέπει να γίνεται μία εκστρατεία πληροφόρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την επόμενη πέμπτη θα έχουμε ένα χρόνο από την ε, λεγόμενη κρίση που οδήγησε σε ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι η κρίση του ψαριού πάγκα, το οποίο έχει μεγάλη διατροφική αξία, αλλά που οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη κρίση ε, πέρυσι και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να έχουμε μια σωστή διατροφή. Αυτές είναι οι βασικές ε, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και που προβάλλω στο πρώτο προσχέδιο. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να μπορέσω να συνεργαστώ με τους σκιώδεις για να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Τόρμον. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, έκθεση, λέει ο κύριος Ντόρμαν, και θα πρέπει να τονίσουμε την κατανάλωση ψαριού που συνεισφέρει στην ε, καλή μας διατροφή και σωστές διατροφικές αξίες. Ε, επίσης πρέπει να συνεργαστούμε με την Νορβηγία, τις νήσους Φερόες και την Ισλανδία. Πολλές φορές πιέζουμε τους προμηθευτές έτσι ώστε να έχουμε τις, την παράδοση και τις παραδόσεις έγκαιρα. Αυτό αφορά και την Ρωσία. Θέλουμε να γίνονται περισσότερες εισαγωγές στην Ευρώπη, αλλά οι εξαγωγείς όπως η Ρωσία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προθεσμίες. Αυτό αφορά και τις καλλιέργειες, την ποιότητα του ύδατος και το γεγονός ότι δεν πρέπει να αμολύνουν το περιβάλλον οι υδατοκαλλιέργειες αυτές. Δεν θα πρέπει να γίνεται πολύ μεγάλη χρήση αντιβιωτικών επίσης στις ε, υδατοκαλλιέργειες και ίσως και καθόλου. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αντιβιωτικά, μόνο όταν είναι απόλυτα αναγκαία. Η κυρία Μίλλε. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Και εμεί ε, θα υποβάλουμε κάποιε τροπολογίε. Γενικώ θεωρώ ότι πρέπει να διαχωρίσουμε μεταξύ τη αύξηση των ε, παραχθησών ε, ποσοτήτων και τη υποστήριξη του υπάρχοντος συστήματο. Αν θέλουμε να αυξήσουμε μόνο του τόνου τη παραγωγή ή αν θέλουμε να δημιουργήσουμε τις περισσότερες θέσεις εργασίας και να διατηρήσουμε τι δομές, είναι σημαντικό να το δούμε. Γι αυτό, η Νορβηγία γι' αυτό είναι επιτυχής, γιατί έχει πολύ συγκεκριμένες και τεχνικές και πολιτικές προϋποθέσεις. οι ε, ε, φάρμες ε, στα Σολομό, πούμε, συνεχώς βρίσκονται υπό επιστημονική παρακολούθηση. Βεβαίως το θέμα του Brexit θα επηρεάσει και την αλία και τη Μεσόγειο για τις θερμοκρασίες του ύδατος, για το βάθος αλίευσης και πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα δούμε γιατί όντως είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Εμείς είμαστε απολύτως υπέρ του να υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση για τους, για πολίτες ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο να δούμε πόσο σημαντικό είναι να καλλιεργεί κανείς ψάρια αλλά βεβαίως πρέπει να δούμε και Ας πούμε, στην ε, ε, Βαβαρία έχουμε πάρα πολλές εκμεταλλεύσεις ε, καλλιέργειας πέστροφας. Πολλές φορές ε, χρησιμοποιείται η θέρμανση από βιοκαύσιμα, ε, μπαίνει η διαδικασία αυτή σε όλη την ε, αλυσίδα και βεβαίως αυτό γίνεται από κοινού με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η, υπάρχουν τα δεδομένα και σε κτηνιατρικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο, έτσι ώστε να αποφεύγονται προβλήματα. Βεβαίως ε, οι κορμοράνοι ας πούμε ή άλλα ε, ε, πτηνά είναι αυτά που αποτελούν ουσιαστικά το βασικό πρόβλημα για την υδατοκαλλιέργεια και όλα αυτά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα ενσωματώσουμε στην έκθεση μέσω τροπολογιών. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπόλαν. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την δουλειά που έκανε για την έκθεση αυτή. Χαίρομαι που δίνουμε έμφαση και στη βιωσιμότητα του τομέα αλλά και στην περιβαλλοντική προστασία και την ασφαλεία των τροφίμων. Ξέρουμε ότι αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα η υδατοκαλλιέργεια ε, και δεν μπορούμε να αφήσουμε το κέρδος αυτό να έρθει εις βάρος της ποιότητας των τροφίμων που καταναλώνουμε. Καταλωσορίζουμε λοιπόν την ανάγκη για περαιτέρω, ευρωπαϊκών, για περαιτέρω ευρωπαϊκές ε, ενημέρωσης για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της ε, βιομηχανίας αυτής. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες ό,τι αφορά την ε, ε, κοινοτική παρέμβαση πριν από την δημιουργία τέτοιων σχεδίων. Ας πούμε στη χώρα μου έχουμε πολυεθνικές οι οποίες δημιουργούν ε, φάρμες τέτοιες ε, ε, στις παράκτητες περιοχές χωρίς όμως καμία συνεννόηση με την τοπική κοινωνία. Πρέπει να υπάρχουν αυστηροί κανόνες για την έκδοση των αδειών λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να, υπάρξει, να αποφύγουμε την, το μονοπόλιο. Και βεβαίω η ευρωπαϊκή πτυχή θα μπορούσε να αποτελέσει και τον θεματοφύλακα, έτσι ώστε να μην καταστρέφονται οι παράκτης περιοχέ όπου δημιουργούνται αυτές οι φάρμες καλλιέργεια. Επίσης, ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο αντίκτυπος που έχει στο περιβάλλον η δεδοκαλλιέργεια σε ό,τι αφορά την ε, μόλυνση, αλλά και την ε, συνύπαρξη με άλλα είδη. Και βεβαίως αυτό εξαρτάται και από το είδος της δεδοκαλλιέργειας. Κάποια είναι πιο επιθετικά, όπως ας πούμε ο Σολομός, κάποια είναι, λίγο, είναι περισσότερο αθώα. Στην Ιλλανδία βλέπετε ποια είναι η, ζημιά που υπάρχει από τα, στα ενδυμικά είδη από την καλλιέργεια σολομού. Οπότε θα θέλαμε να υπάρξει μια, ένας καθορισμός προτεραιοτήτων για την προστασία των ενδικών, ενδυμικών ε, ειδών ε, σε σχέση με τα ε, είδη που καλλιεργούνται στις φάρμες για να μπορέσουμε έτσι να μειώσουμε και τον, αντίκτυπο στο, τον περιφυλακτικό αντίκτυπο και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και τα χωροκατακτητικά είδη. Ευχαριστώ you. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Έξτον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για την γνωμοδότησή του. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και χαίρομαι πολύ που συνεργάστηκα μαζί του. Καταρχά να πω ότι δεν συμφωνούμε απολύτω με την πρώτη παράγραφο του σχεδίου γνωμοδότηση που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει την παραγωγή στην, ε, το, στον τομέα τη εντατοκαλλιέργεια, λαμβάνοντα υπόψη την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τι περιβαλλοντικέ πτυχέ. Θα θέλαμε η βιώσιμη και περιβαλλοντικά στερεή υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να αποτελεί το, την, προ, προϋπόθεση για να αυξηθεί η, η παραγωγή. Επίσης, η αυξανόμενη παραγωγή υδατοκαλλιέργειας προτείνεται ως αναγκαιότητα για να επιτευχθούν οι ανάγκες σε ψάρια του πληθυσμού μια βασική προτεραιότητα για να καλύψουμε την αυξανόμενη ανάγκη είναι ε, ο εμπλουτισμό, ο επανεμπλουτισμό των ε, εχθιακών αποθεμάτων. Επίση, η βιωσιμότητα της, ε, του τομέα τη ειδοκαλλιέργεια πρέπει να προωθηθεί μέσω βιώσιμου παγκοσμίου εμπορίου, με διατάξει για το πώ θα τηρούνται τα περιβαλλοντικά πρότυπα στι συμφωνίε Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε και τι δικές τους, τους δικού του κλάδου ειδοκαλλιέργεια. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η υδατοκαλλιέργεια της θα πρέπει να είναι βιώσιμες, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει ως εξή. Να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη επαρκούν, επαρκούς ζωοτροφής, θεοτροφής για τα ψάρια. Η μείωση της, του αντικτύπου στην βιοκαλλιέργεια και η, χρήση, η, λιγότερη, η μικρότερη χρήση χημικών. Για, τις, για τα ηχθιάλευρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ε, ηχθιαλέων και ηχθιαλεύρων ε, ε, βιώσιμης παραγωγής και βεβαίως θα πρέπει σε περιβαλλοντικό επίπεδο αυτό όλο να είναι ανεκτό. Οι τεχνολογίες που υπάρχουν θα πρέπει να αποτελέσουν προϋπόθεση για την καλύτερο έλεγχο και ανιχνευσιμότητα έτσι ώστε να αποφύγουμε προβλήματα ο αντίκτυπο ε, και τα ωφέλη τη ε, της για τα διάφορα είδη στη διαφύλαξη τη ε, βιοπικιλότητα σημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω έρευνα για να δούμε ποιο αντίκτυπο υπάρχει από την δεδοκαλλιέργεια στα ενδημικά είδη. Θα πρέπει να υπάρξει ένα τοπικό σχεδιασμό, κάποιοι περιορισμοί, για τις διάφορες ζώνες που θα τεθούν ως ζώνες υδατοκαλλιέργειας και επίσης η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να ενθαρρύνει την υδατοκαλλιέργεια μέσω περιβαλλοντικών υπηρεσιών και ε, ε, επέκταση των ζωνών αλίευσης, ε, να υπάρχουν και κάποιες κάποιες ίσως ψυχαγωγικές περιοχές που θα μειώσουν τον ατροφισμό. Υπάρχει και η υδατοκαλλιέργεια RES ενός συστήματος επανακυκλοφορίας που χρησιμοποιεί δηλαδή το ε, νερό το οποίο την χάνει χημικής επεξεργασίας αλλά βεβαίως το θέμα των ηχθειοτροφών ε, παραμένει. Δεν μπορεί αυτό να είναι βιώσιμο εάν δεν λύσουμε πρώτα το προηγούμενο πρόβλημα. Τέλος, να μειώσουμε τον ε, αντίκτυπο της χρήσης χημικών. Η χρήση χημικών και αντιβιωτικών ε, δημιουργεί προβλήματα στα οικοσυστήματα αλλά και στην ανθρώπινη υγεία. Η ομάδα μου πιστεύει ότι τα τοξικά χημικά και τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται στι χιστιοτροπέ θα πρέπει να αντικατασταθούν από πιο ασφαλεί εναλλακτικέ. Θα υποβάλουμε κάποιε τροπολογίε για τα θέματα αυτά και βεβαίω προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η γνωμοδότηση και την υδατοκαλλιέργεια θα είναι αυτή που θα θέτει ω προτεραιότητα το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων και την ε, παραγωγή των ηχθείων. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, ο κύριος Λάινεμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ε, ευκαιρία να αντιδράσω. Πριν από κανένα χρόνο, ο Επίτροπος Βέλα έκανε μία ερώτηση στην, στον μηχανισμό επιστημονικής συμβουλής ε, της Κομισιόν πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερη βιομάζα από τους ωκεανούς και να έχουμε παράλληλα βιώσιμη διαχείριση. Η ομάδα αυτή, ε, όπως περιμένετε, απάντησε ότι θα πρέπει να έχουμε βιώσιμη ε, αλλά και η χθιοκαλλιέργεια θα πρέπει με βιώσιμο τρόπο να παράγει περισσότερη ε, τροφή στο παρελθόν για να καλύψουμε και τις ανάγκες των 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που θα έχουμε στο μέλλον, ε, διατηρώντας και, το, και τη ζωή στους ωκεανούς μας. Αυτή είναι μια κατευθυντήρια γραμμή. Μέσα σε αυτή θα πρέπει να πορευτούμε για να διατηρήσουμε την, ε, μια υψηλή ποιότητα ε, ηχθειοκαλλιέργεια, ε, με υψηλά πρότυπα που ούτω ή άλλω είναι τα υψηλότερα σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και με του ενδιαφερόμενου για να εξαλειφθούν οι φραγμοί για να, που παρεμποδίζουν την ε, γιγάντωση του τομέα. Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να βελτιωθούν, δεν πρέπει να υπάρχει ε, διοικητικό άχθος. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε πού μπορεί η εκμετάλλευση αυτή να εγκατασταθεί καλύτερα, στη θάλασσα ή στην ξηρά. Ε, θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό ο τομέα και ισοτιμία σε σχέση με τις εισαγωγές. Αυτή η πολιτική έχει και την υδατοκαλλιέργεια γλυκού νερού που ανεφέρθηκε από μια Ευρωβουλευτή. Υπάρχουν κάποια καλά νέα. Μετά από χρόνια υπάρχει μία αύξηση μεταξύ του 2014 και του 2015 με βάση τα τελευταία στοιχεία, γιατί τότε τα έχουμε, από μάλλον κατά 4% ε, κατόγκο και 8% ε, σε οικονομικό μεγέθη. Εφτάσαμε φτάσαμε στα, σε 3 εκατομμύρια τόνους. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει νόμους ε, που αφορούν ειδικά την ηχθειοκαλλιέργεια και διευκολύνουν την αδειοδότηση. Έχουν θαλάσσια ε, σχέδια σχεδιασμού και έχουν ειδικέ δομέ για τη διαχείριση του περιβάλλοντο. Τώρα κάνουμε μια διάμεση αξιολόγηση τη ανοιχτή μεθόδου συντονισμού που είναι η της τη Κομισιόν για να προωθήσει την ηχθειοκαλλιέργεια. Η ανάγκη για μια εκστρατεία αναφέρθηκε. Έχουμε μια εκστρατεία που λέγεται ε, καλλιέργεια στην Ευρώπη εδώ και χρόνια και είναι ε, λαμβάνει υπόψη το, τις ανάγκες ε, κάθε κράτους μέλους. Ε, η Ιρλανδία και η Κροατία ε, θα είναι στο κέντρο αυτής της εκστρατείας φέτος. Φυσικά αυτό δεν αρκεί. Την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, οργανώνουμε ένα σεμινάριο στην Επιτροπή των Περιφερειών, μαζί με την Επιτροπή των Περιφερειών, για να τονώσουμε, τονίσουμε μάλλον τη σημασία των περιφερειών στην ηθιοκαλλιέργεια. Γιατί ορισμένες παρεμβάσεις αναφέρονται την ε, τοπική ανάπτυξη, που είναι σημαντικό τμήμα τη ηχθειοκαλλιέργεια. Να είναι πιο κοντά η ηχθειοκαλλιέργεια στου τοπικού πληθυσμού. Υπάρχουν καλά παραδείγματα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλία ε, βοηθάει τι τοπικέ κοινότητε μέσω α, ομάδων α, δράσεων για τις τοπικές ε, κοινωνίες. Και στη Γερμανία, στο Κάπεν, που έχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα που ε, εδώ και χίλια χρόνια διατηρούν και το φυσικό αλλά και το τεχνητό περιβάλλον, ε, μας δίνει ε, μία περίπτωση καλού παραδείγματος, ας πούμε. Επίσης, τελευταίο, σημαντικό, η ανάγκη για επενδύσεις. Ε, αναφέρθηκε ότι είναι κλειστό κύκλωμα. Ε, υποστηρίζουμε με έρευνα αλλά και με άμεση χρηματοδότηση τις καινοτόμες προσεγγίσεις που μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε την, τα ψάρια μας. Ε, μπορούν να υπάρχουν μοντέλα για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ποιότητα. Ε, επίσης, ε, υπάρχουν μοντέλα τα οποία δεν θέλουν τόσο πολύ νερό ε, για να χρησιμοποιηθούν από χώρε που υπάρχει η έλλειψη νερού. Επίσης δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο το ψάρι και τα καρκινοειδή, ε, τα μύδια κτλ. αλλά και τα φύκια, τα μικροφύκια ε, και το περιβάλλον, δηλαδή το θαλάσσιο, ε, θαλάσσιο περιβάλλον. Υπάρχει ένα φόρουμ για το θαλάσσιο περιβάλλον, βιολογικό θαλάσσιο περιβάλλον, ε, για να δούμε πώς μπορούμε να παντρεύσουμε τα δύο, την οικονομία, ας πούμε, το περιβάλλον. Επίσης, υπάρχει ένα, μια πλατφόρμα επενδύσεων για την μπλε οικονομία, ούτως ώστε να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις στον τομέα. Ε, και αυτά. Καιρός να σταματήσω πια. Thank you. Now I will give the floor to the rapporteur. Συγητής, ο κύριος Γκαμπούς, για να ολοκληρώσει. Μάλιστα. Πολύ σύντομα. Να ευχαριστήσω όλες όλου του ομιλητέ για τι παρεμβάσει. Έχουμε ένα κοινό παρανομαστή, νομίζω, το οποίο, ο οποίο συνοψίζεται στο εξή. Ότι το θέμα είναι σημαντικό. Θα πρέπει να εστιάσουμε την πολιτική ηχθειοκαλλιέργεια με ένα τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να μην ξεχνάμε την επίπτωση που έχει στον τοπικό πληθυσμό. Και φυσικά, η πολιτική ηχθειοκαλλιέργεια θα πρέπει να συνδέεται με την έννοια της βιωσιμότητας, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και την έννοια της ποιότητας και με την έννοια της α, κυκλικής οικονομίας. Ε, η παραγωγή, θα, τοπική παραγωγή ε, έχει να κάνει με την εγκύτητα που έχει με τις α, τοπικές αρχές και τοπικές δομές. Εγώ δεν θέλω να μιλήσουμε για παραγωγή με βάση επιχειρηματικά κριτήρια. Ε, είναι το σχήμα. Μην ξεχνάτε ότι πέρα από αυτό υπάρχει και το θέμα των ωκεανών που πρέπει να διαχειριστούμε με πιο βιώσιμο τρόπο και πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Τώρα, για την ηχθειοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, γλυκού νερού, συμφωνώ απολύτως με την υποσημείωση της κυρίας Μιουλέρ. Και εμένα ως εισηγητή μου συνέβη αυτό που συνέβη σε... όταν ένας, μεσογεία... όταν ένας ε, νότιος ας πούμε πηγαίνει αλλού, σε μια άλλη χώρα. Ε, μερικές φορές οι Βόρειοι ξεχνάνε ας πούμε ότι και τα δικά μας δάση καίγονται, αλλά και εμείς ξεχνάμε ας πούμε ότι υπάρχει υδατοκαλλιέργεια και ηχθειοκαλλιέργεια γλυκού νερού σε άλλες χώρες ας πούμε που είναι μακριά από τη θάλασσα. Ε, Κάνουμε τέτοια λάθη. Ε, δεν, θα, δεν το κάνω αυτό το λάθο. δεν θα το ξεχάσω, δεν θα ξεχάσω και, τις, και ε, την ηχθειοκαλλιέργεια του γλυκού νερού την ώρα που θα βελτιώσω πούμε, την, το κείμενό μου. Και θα λάβω υπόψη μου βεβαίω και τι τροπολογίε και θα έρθω σε επαφή με του κοιόδη συζητητέ για να τι δουλέψουμε μαζί. Ε, η νέα ε, προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 11 η ώρα 31 Ιανουαρίου. Το επόμενο σημείο είναι αυτό που θα μας απασχολήσει τώρα αλλά στις 11 και 4 έχουμε τον Βούλγαρο Υπουργό. Η εφαρμογή της ΚΑΠ για τους νέους αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη μεταρρύθμιση του 2013. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε χρόνο, το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν ε, μπορώ να σας πω ότι είναι έξι η παραγραφή της έκθεσής μου. Ε, χρειαζόμαστε μια νέα γενιά ε, αγροτών, το ξέρω, είναι δύσκολο να το πετύχουμε σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά το βασικό είναι να έχουμε περισσότερους νέους ε, γεωργούς. Και σε αυτή την έκθεση εξετάζουμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η ΚΑΠ αφορά τις ανάγκες των νέων ε, γεωργών. Θέλουμε οι νέοι αυτοί να έχουν ε, τα περιβαλλοντικά, τις περιβαλλοντικές τεχνικές γνώσεις για να υποστηρίξουν μια βιώσιμη γεωργία. Επομένως η κατάρτιση και τα προσόντα είναι σημαντικά και υπάρχει και μια βασική προσέγγιση ε, παράγραφος ή παράγραφος 5, όπου μιλάμε για την ανάγκη ε, συνοχής ανάμεσα στην ευρωπαϊκή διάσταση και στην δράση των κρατών μελών. Ε, σε ό,τι αφορά τους νόμους διαδοχής, κληρονομιάς δηλαδή, και φορολογίας, Ούτω ώστε να υπάρχει ανανέωση στις γενιές των γεωργών και να περνάει ας πούμε, η γεωργική εκμετάλλευση από τη μια γενιά στην άλλη. Πολύ σημαντικό αυτό. Και τελευταία παράγραφος στην έκθεση μιλάει για μια ολιστική προσέγγιση για να διευκολύνει την πρόσβαση στην γη για τους νέους γεωργούς, αλλά και για να τους δώσει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, σε υπηρεσίες συμβουλευτικές και συμβουλευτικά συστήματα, αλλά και εκεί που ζουν θα πρέπει να έχουν τις ίδιες υπηρεσίες με τους νεαρούς ε, ομολόγους τους που ζουν στις πόλεις. Ε, να πρέπει να έχουν ευρεία ζώνη, υπάρχει ευρυζωνικότητα δηλαδή και υγειονομικές υπηρεσίες. Είμαι ανοιχτή στα σχόλια το των συναδέλφων είναι η άγκρη καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Πάντως είναι σημαντική αυτή η έκθεση, είναι προτεραιότητα για την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Κλείνω με αυτά τις παρατηρήσεις μου και περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων. very much. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τζεντήλε. Εντάχει, Πρόεδρε, το θέμα είναι αποφασιστική σημασίας αν σκεφτούμε την Ευρώπη που θέλει να αναπτυχθεί, να ε, ευημερεί και να έχει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μιλάμε για την έννοια της ε, αγροτικής επιχείρησης που θα πρέπει να προαχθεί έτσι ώστε χιλιάδες νέων να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό το νέο επαγγελματικό και οικονομικό πλαίσιο και να μπορέσουν να ε, δράσουν αυτόνομα Πιστεύω ότι και η Ευρώπη μπορεί να χτίσει γύρω από αυτή την ιδέα και ιδιαίτερα αυτή την ανάγκη κατάρτισης και ιδιαίτερα επαγγελματικής κατάρτισης γιατί η γεωργία είναι όλο ένα και πιο ε, τεχνολογικά ανώτερη αλλά και καινοτόμα. Γιατί κανείς θα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται την επιχείρησή του και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσαρμοστεί κάπου μέσα στα πλαίσια των διατάξεων Omnibus και να προβάλλει μέσα τα οποία θα μπορέσουν να αποσοβήσουν τους κλειδονισμούς του συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν να χτίσουμε αυτές τις νέες αρμοδιότητες και διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα για να βοηθήσουμε τους αγρότες ε, να μπορέσουν να γίνουν και γεωκτήμονες ε, έτσι ώστε να αποφύγουμε τη, τα προσκόμματα του παρελθόντος, να μιλάμε για μια σύγχρονη προσέγγιση όπου θα συμμετέχουν ε, περισσότεροι εμπλεκόμενοι φορείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Μαγκίνες ε, για αυτή τη γνωμοδότηση. Πράγματι υπάρχουν ε, ένα και περισσότερες ανισότητες μεταξύ υπαίθρου και αστικών κέντρων. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε συνεπείς, θα πρέπει κάπως να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα θα πρέπει να εγγυηθούμε ώστε οι αγροτικές περιοχές και οι γεωργοί να μην αποχωρήσουν από τις αγροτικές περιοχές, να μην γίνει δηλαδή απερίμωση το, της υπαίθρου. Θα πρέπει οι νέοι να χρησιμοποιούν όλο ένα και περισσότερη τεχνολογία και περισσότερο την τεχνολογία και θα πρέπει να πείσουμε τους νέους για το μέλλον της αγροτικής οικονομίας. Είτε ζουν στην Ήπεθρο είτε στις κομοπόλεις. Δηλαδή το περιβάλλον δεν αρκεί. Θα πρέπει να έχουμε να έχουν και πρόσβαση σε ευρυζωνικά συστήματα. Θα πρέπει να υπάρχουν κοινά συστήματα κανόνων έτσι ώστε να μην, Thank να μην προστίθενται προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα. Η κυρία ακόμα ...31,5% είναι ε, αγρότες γύρω στα 65 ε, έτη. Οι βασικές αιτίες λοιπόν του προβλήματος είναι ότι ε, πρέπει να δούμε πιο ε, οικονομικά, ε, οικονομικούς όρους για, την, για το δανεισμό των των αγροτών και επίσης το θέμα της κοινωνική ασφάλισης τους. Αυτά τα δύο θέματα νομίζω ότι πρέπει να τα συμπεριλάβουμε ε, στο κείμενο. Είναι σημαντικό επίσης η νέα, ε, η, ε, η νέα γενιά να έχει την ευκαιρία να προσφέρει τις δικές της ιδέες, απόψεις, μεθόδους για την γεωργία για πολλούς μεγαλύτερης ηλικία ε, βεβαίως αυτό ίσως να θεωρείται ε, ως απώλεια η μείωση και θεωρούν ότι είναι ε, πρόβλημα. Αυτό το εμπόδιο λοιπόν θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως η περαιτέρω εκπαίδευση των γεωργών είναι σημαντική. θα πρέπει όντως να δούμε την όρεξη να γίνει κανείς ε, ε, γεωργός κάτι ε, θετικό για το επάγγελμα του Γιώργου, έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε ένα θετικό image αυτού του επαγγέλματος. Αν όταν έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση βέβαια το image συνήθως είναι θετικό. ευχαριστώ και την εισηγήτρια και βεβαίως κάποιες τροπολογίες θα υποβάλω κι εγώ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω εγώ την κυρία Μαγκίνες. Ουσιαστικά τους ε, νέους γεωργούς μπορούμε να τους προσφέρουμε την δυνατότητα να δουλέψουν όταν μπορούμε να τους εγγυηθούμε και ένα εισόδημα το οποίο θα τους βοηθά να ζήσουν. Γι' αυτό οι ε, προοπτικές βεβαίως τώρα δεν είναι πάρα πολύ καλές. Το εισόδημα των ε, γεωργών κυρίως για τις μικρές εκμεταλλεύσεις είναι περίπου το μισό ε, σε σχέση με άλλους τομείς και από εκεί νομίζω εξαρτάται για να δώσουμε προοπτικές στους νέους και σε ό,τι αφορά το αύξηση του εισοδήματο, αλλά και γενικώ μακροπρόθεσμε προοπτικές και ε, να μπορεί κανείς δηλαδή να ζήσει στην ε, Ήπεθρο με το εισόδημα που θα έχει. Οι υποδομές θα πρέπει να είναι ε, βελτιωμένες και όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα δούμε από κοινού με τη γεωργική πολιτική και την ανάπτυξη υπέρθρου. Αν θέλουμε να έχουμε αρκετούς νέους γεωργούς, τότε ουσιαστικά το θέμα είναι η εκπαίδευσή τους και ίσως εδώ να μην έχουμε απόλυτα σωστή προοπτική. Θα πρέπει να ε, τονίσουμε το θέμα της βιωσιμότητας, της βιολογικής καλλιέργειας, αλλά και την θέση σε εμπορία. Νομίζω ότι έχουμε επικεντρωθεί πολύ στις μεθόδους παραγωγής και λίγο στο πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε την ιδέα του να είναι κανείς γεωργός επαγγελματικά. Ε, κάτι που είπε επίσης η κυρία Μαγκίνες είναι το πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στο ε, επάγγελμα. Οι ε, τιμές για να αποκτήσει κανείς γη είναι πολύ υψηλές πια. Και βεβαίως πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα προγράμματα δανεισμού. Πολλές φορές ε, λόγω αυτού δεν μπορούν να φτάσουν καν στην απόκτηση γης οι γεωργοί. Και ένα τελευταίο σημείο. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να, το, να βάλουμε κάποιο όριο ηλικίας εδώ. Νομίζω ότι όλοι όσοι θέλουν να μπουν στον κλάδο να έχουν την ευκαιρία. Μπορεί κάποιο να θέλει στα 45 του, α πούμε, να γίνει γεωργό. Δεν θα πρέπει να του βάλουμε όριο και να του πούμε όχι. Όλοι όσοι θέλουν να μπουν στον κλάδο θα αποτελέσουν κέρδο για τον κλάδο τη γεωργία. Οπότε εγώ υποστηρίζω την έκθεση και βεβαίω θα υποβάλουμε και εμεί κάποιε παρατηρήσει για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον τη γεωργία. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή στον κύριο Βάσκο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση και τη συνεισφορά της Επιτροπής σας γενικά που θα οριστικοποιηθεί και με την συνεργασία της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Στις 29 Νοεμβρίου ε, συντάξαμε μία ανακοίνωση για την ε, καλλιέργεια των γεών και την αγροτική οικονομία. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους αγρότες και αυτό είναι ύψης της σημασίας για την ΚΑΠ και για το μέλλον της ΚΑΠ. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μετάβαση σε μία βιώσιμη και καινοτόμα γεωργία. Και αυτό σημαίνει και ανανέωση του ανθρωπίνου δυναμικού, δηλαδή θα γίνει η μετάβαση της γνώσης έτσι ώστε η γνώση η οποία γεννάται και προκύπτει να οδηγήσει σε μία πιο βιώσιμη γεωργία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προτρέψουμε περισσότερους νέους στις αγροτικές δραστηριότητες. Και βλέπουμε ότι οι νέοι γεωργοί ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο να θέσουν σε εφαρμογή νέες τεχνολογίες που να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και νομίζουμε ότι αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να διαχωριστούν. Γι' αυτό αυτό. Είναι πολύ θετικό το ότι σας απασχόλησε αυτό το θέμα. Τώρα, δύο ειδικά σημεία. Στην ΚΑΠ ήδη έχουμε μία εργαλειοθήκη για να υποστηρίξουμε τους νέους γεωργούς. Υπάρχει όμως η, ικανότητα να γίνουν αυτά τα μέσα πιο αποτελεσματικά και γι' αυτό υποστηρίζουμε και προσμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικέ ανάγκες των νέων. Και ένα άλλο στοιχείο που αντικατοπτρίζεται στην έκθεση και στην ανακοίνωσή μας είναι το εξής. Πέρα από τις ε, κοινέ μας προσπάθειες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία ε, αποφασίζουν σε επίπεδο κρατών μελών για ιδιαίτερα ως προς την ε, χρήση των γεών, κληρονομιά γεών και φορολόγησή τους και πολλές φορές δημιουργούνται εμπόδια για να μπει κανείς στο, στην οικονομία αυτή, ιδιαίτερα όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή μας, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνοχή του τι κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι γίνεται σε εθνικό. Πιστεύουμε ότι η γενική προσέγγιση για τη μελλοντική ΚΑΠ θα κινείται προς ένα σύστημα στοχοθέτησης για να βοηθήσουμε τις αγροτικές κοινότητες, βεβαίως αναγνωρίζοντας την επικουρικότητα και τον ρόλο των κρατών μελών που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της επικράτειας. Αυτό το πρότυπο θα ήταν πολύ καλό για την αναγέννηση του τομέα για να ε, αντιμετωπίσουμε και την τροχοπέδη εισόδου σε αυτό το τομέα. Η κυρία Μαγκίνες, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα πολύ επικοδομητικά σχόλια. Νομίζω σε αυτά που είπε ο κύριος Χόισλινγκ ε, έχει απόλυτο δίκιο, αλλά η πρώτη παράγραφος ασχολείται με αυτά τα θέματα, με το θέμα της βιωσιμότητας, αλλά δέχομαι βεβαίως τροπολογίες. Ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να διαφωτιστεί αφορά τους νέους, ε, αλλά κυρίως γυναίκες, τις νέες γυναίκες στην Ιρλανδία ε, υπάρχει μία ομάδα γυναικών που θα συναντηθεί σήμερα για να δει το μέλλον της στον τομέα της γεωργίας. Και από αυτό τον ε, διάλογο με τους γεωργούς βλέπω ότι οι νέοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες, να δουν την περιβαλλοντική διάσταση και γι' αυτό οι γυναίκες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτή την πρόπτικη. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα αμετακίνητο σύστημα βοήθειας, γιατί πολλοί χάνουν από αυτό το σύστημα. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον της ΚΑΠ, βρέθηκα σε μία τεχνική συνεδρίαση ε, γύρω από την ανακοίνωση της Επιτροπής και θα ήθελα οι συνάδελφοι να το κοιτάξουν εις βάθος, γιατί τώρα που κατανοώ καλύτερα το ζήτημα, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει τόσο η συμμόρφωση, αλλά τα αποτελέσματα, δηλαδή θα πρέπει να τονίζουμε στους γεωργούς τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν, όχι τι δεν μπορούν να κάνουν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευελιξία σε επίπεδο κρατών μελών για να δουν κατά πόσο πρέπει να κάνουν περισσότερα για νέους. Και θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται η διασύνδεση μέσων σε εθνικό επίπεδο. Αναμένω τι τροπολογίε σας μέχρι την επόμενη Πέμπτη στις 12, όπως θα το επιβεβαιώσετε και εσείς και θα χαρώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους, θα συναντηθούμε με τους σκιώδη σύντομα. Η προθεσμία είναι η 3η Φεβρουαρίου στις 11 η ώρα το μεσημέρι. Μπορούμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Υπουργό Υγείας, Mm, yes. Uh, let me say hello to the minister. τον Υπουργό. Καλώς ήρθατε. Με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε αυτή τη συζήτηση και θα σας δώσω το λόγο πάρα αυτά. Ευχαριστώ. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας που έχετε στις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τιμή μου να παρουσιάσω το πρόγραμμά μου στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, την Επιτροπή ΕΜΒΗ. Ε, που είναι υπεύθυνη για το περιβάλλον, ε, δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων. Η Βουλγαρία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μελλοντικέ εξελίξει Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτώνται από τι ε, συζητήσει και το αποτέλεσμα των συζητήσεων του επόμενου μήνε. Για να μπορέσουμε να επιλέξουμε το σωστό τρόπο, θα πρέπει όλοι μαζί να καταγράψουμε τις προκλήσεις, τα επιτεύγματα και τα λάθη, ούτως ώστε να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά για να το κάνουμε πρέπει να είμαστε μαζί. Για τη Βουλγαρία είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την ενότητά τη. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να μείνει ενωμένη και δυνατή. Εμείς ως Προεδρία πιστεύουμε ότι όταν είμαστε μαζί είμαστε δυνατοί. Η προσέγγιση μας είναι συνένεση, συμβιβασμός και συνεργασία. Είμαστε υπέρ μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η οικονομική ανάπτυξη είναι ένα εργαλείο για να πετύχουμε κοινωνική ισότητα και ευημερία για τους πολίτες όλων των κρατών μελών. Θα δουλέψουμε για μια Ευρώπη ασφαλή, σταθερή και αλληλέγγυα και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ειρήνη για τους λαούς μας και τους γειτονές μας. Είμαι εδώ σήμερα για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες στον τομέα της υγείας και να απαντήσω οπωσδήποτε στις ερωτήσεις σας. Τους επόμενους μήνες θα γίνουν συζητήσεις για τη μελλοντική χρηματοδότηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μέλλον των βασικών τομέων συνεργασίας. Πιστεύω ότι μια ενωμένη Ευρώπη είναι αδιανόητη χωρίς βασικές αξίες όπως η υγεία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Ανεξάρτητα από τις διαφορές μεταξύ των συστημάτων των κρατών μελών, η συνεργασία σε αυτού του τομεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς ανάγκη να περάσουμε στην αρμόνιση, δίνει απτά ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες σε καθημερινή βάση. Ποιοι είναι οι τομείς υγεία όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής έχει κάνει κάποια πράγματα με δραστήρια πολιτικά μηνύματα, πρωτοβουλίε και νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για την ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών σε όλη την Ευρώπη. Είναι η οδηγία του 2011, υπαριθμών 24, για την ε, εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγεία. Εδώ βασιζόμαστε και σε ηλεκτρονικές λύσεις άμα χρειαστεί. Με την ενεργή υποστήριξη της Κομισιόν υπάρχει ένα δίκτυο ε, υψηλής, υψηλά εξειδικευμένων κέντρων ε, αγωγής και θεραπείας, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς ε, και με την ε, πραγματογνωμοσύνη όλων των εθνικών ε, υπηρεσιών φαρμάκων και το συντονισμό από, την Ευρωπαϊκή, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον ΕΜΑ, ε, προσπαθούμε να δρομολογήσουμε ε, καινοτόμα φάρμακα ψηλής ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας και να εξασφαλίσουμε την ε, φαρμακοεπαγρύπνηση, κανονισμό 726 κάθος 2004 και να εφαρμόσουμε όλο το πλαίσιο νομοθεσίας με τις οδηγίες, κανονισμού ε, για τα παιδιατρικά φάρμακα, τα ορφανά φάρμακα κτλ. Έχουμε λεπτομερείς κανονισμούς για την ε, θέση στην αγορά και την αδειοδότηση φαρμακευτικών προϊόντων για κλινικές δοκιμές, κανονισμός 536 του 2004 για τις ιατρικές συσκευές και συσκευές για διάγνωση in vitro, κανονισμός 2017-745 και 2017-746. Υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τα, τους ιστούς, τα όργανα και τα κύτταρα, για τη δωρεά οργάνων και, ε, και τη μεταμόσχευση. Υπάρχουν ευκαιρίες στην εσωτερική αγορά για την ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών και γιατρών και την ανταλλαγή εμπειριών. Ένας μηχανισμός για κοινή συντονισμένη απόκριση από όλα τα κράτη-μέλη και αυτό έχει δημιουργηθεί για να ελέγξουμε την διάδοση μεταδοτικών ασθενειών και τι διασυνοριακέ απειλέ υγείας. Αυτοί οι μηχανισμοί βασίζονται και θα συνεχίσουν να βασίζονται στην εθνική πραγματογνωμοσύνη. Ακριβώς γι' αυτό είναι σημαντικό αυτή η πραγματογνωμοσύνη να προωθηθεί και να απτυχθεί σε όλα τα κράτη-μέλη και να υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι ο τρόπο για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του συστήματος υγείας, μάλλον των συστημάτων υγείας. Διάφορα πολιτικά έγγραφα, συμπεράσματα του Συμβουλίου, ε, ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίζουν τη σημασία των πολιτικών για τις μεταδοτικές και μη μεταδοτικές χρόνιες ασθένειες, δραστηριότητες για την πρόληψη των ε, ασθενειών που εμφανίζονται όπως ε, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές αρρώστιες. Το να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους όπως το αλκοόλ, ο καπνός, ε, και η μη υγιεινή διατροφή απαιτεί συντονισμένο επίπεδο και προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην Υγεία, όλα τα πολιτικά μηνύματα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και στις συστάσεις του Συμβουλίου, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνουν μια έντονη όθηση στις πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ σημαντικές γιατί είναι η ευκαιρία για να ανταλλάξουμε εμπειρίε και βέλτιστες πρακτικές, να μάθουμε ένα από τον άλλον, βλέποντας τι πραγματογνωμοσύνη έχει το κάθε κράτος μέλος και συνενώνοντα αυτή την γνώση και μαθαίνοντας για τα μοντέλα υγείας και τις καλέ πρακτικές που έχουν οι άλλοι. Το πολιετές πρόγραμμα υγείας συνεισφέρει σημαντικά σε αυτή τη συνεργασία. Έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο γιατί υποστηρίζει πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας. Η εφαρμογή κάθε πρωτοβουλία και νομική πράξη και νομοθετικού κειμένου, καθώ και των ευρωπαϊκών, απαιτεί ότι αυτοί που εφαρμόζουν αυτά τα κείμενα δεν είναι όμως, δεν είναι απλό τμήμα της διαδικασίας για το σχεδιασμό, αλλά έχουν και έναν ηγετικό ρόλο να παίξουν εν συνεχεία. Η υγειονομική περίθαλψη είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που είναι η πιο απτή από οποιαδήποτε άλλη για τη ζωή των ανθρώπων. Ε, η Ευρώπη θέλει να πετύχει περισσότερη ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Οι πρωτοβουλίε στην τομέα τη υγεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχουν σαν στόχο όχι μόνο να υποστηρίξουν τη βιομηχανία και την καινοτομία, αλλά πάνω απ' όλα την ανάγκη προστασία ανθρώπινη υγεία. Ό,τι προϊόν και να υπάρχει στην αγορά, φάρμακα, τρόφιμα κτλ. Όποια και αν είναι αυτά, πάνω απ' όλα πρέπει να, είμαστε, να έχουμε γνώση για τι και επίγνωση για τι επιπτώσει στην ανθρώπινη υγεία. Αλλιώ κινδυνεύουμε να χάσουμε το πιο πολύτιμο πράγμα, την εμπιστοσύνη του κόσμου στο σύστημα. Να υπενθυμίσω ότι είναι ανάγκη για να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασία υγεία υπάρχει και στι συνθήκε. Στην ε, συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 114, όταν προωθούνται πρωτοβουλίες εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτή η υποχρέωση μας βαραίνει όλους, την Κομισιόν, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτό είναι ακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουμε σχεδιάσει και προγραμματίσει τις προτεραιότητές μας στον τομέα της υγείας ως Προεδρία. Το κάναμε γνωρίζοντας ποιο είναι το πλαίσιο, γνωρίζοντας ότι θα είμαστε και στο τιμόνι των συζητήσεων για τους επόμενους 6 μήνες. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα δώσουμε προτεραιότητα σε δύο πολιτικά σημαντικά θέματα υγιεινή διατροφή για τα παιδιά και την ανάγκη για αποτελεσματικά φαρμακευτικά προϊόντα σε καλές τιμές, προσιτές τιμές. Υγιεινή διατροφή για τα παιδιά. Αυτό είναι ένα θέμα τεράστιας σημασίας. Ένα θέμα που συνδέεται με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Το μέλλον μιας ανταγωνιστικής Ευρώπης είναι αδιανόητο χωρίς μια υγιεινή ε, υγιή και με καλές εκπαιδευτικές βάσεις νέα γενιά. Η προοπτική στο θέμα της υγείας ε, έγκυται στην διατροφή που κάνουν τα παιδιά, γιατί είναι βασικό στοιχείο της υγείας των παιδιών. Η μη υγιεινή διατροφή ε, εξαπλώνει ε, και διαδίδει χρόνιες αρρώστιες στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έχουμε σχεδιάσει συζητήσεις για την επίπτωση των διατροφικών συνηθιών την υγεία των παιδιών ε, στη φυσική και διανοητική τους ανάπτυξη. Θα συζητήσουμε για την ανάγκη ε, τροφίμων που να μην είναι απλώς ασφαλή, αλλά υγιεινά ε, η θέση στην αγορά των τροφίμων. Και την ανάγκη να διατηρήσουμε τις παραδοσιακές διατροφές στην Ευρώπη και την ανάγκη να διατηρήσουμε την πολυμορφία. Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε υγιή παιδιά και υγιή πληθυσμό και εργατικά χέρια. Αυτή η συζήτηση θα ενισχύσει και θα τροφοδοτήσει και τις συζητήσεις για την κοινή γεωργική πολιτική και το μέλλον της. Η επιτυχία των πολιτικών πρόληψης εξαρτάται από την διαθεσιμότητα στην αγορά τροφίμων που είναι και υγιεινά και σε προσιτές τιμές η υγεία και η γεωργία ε, θα πρέπει να συνεργάζονται με αυτές, σε αυτές τις προτεραιότητες. Στις 6 Φεβρουαρίου στη Σόφια ε, θα γίνει μια συζήτηση εμπειρογνωμόνων και θα γίνουν και συζητήσεις στο Συμβούλιο για τα συμπράσματα του Συμβουλίου ε, τον, στις 22 Ιουνίου. Επίσης, ένα άλλο όλο και πιο επίκαιρο θέμα είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα. Ε, θέλουμε να δούμε το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η θεραπεία που προσφέρουν και αν υπάρχει καλή σχέση ε, κόστους-οφέλους, ε, γιατί μιλάμε για το δημόσιο χρήμα. Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο υποστηρίζει την καινοτομία, εξασφαλίζοντας και την ασφάλεια των ασθενών. Να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία είναι προϋπόθεση για να υπάρχει εμπιστοσύνη από πλευρά ασθενών. Γι' αυτό ακριβώς η προοπτική της υγείας θα πρέπει να είναι ε, στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων που κάνουμε για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Είναι απαράδεκτο η αγορά και ειδικά η ευρωπαϊκή ε, ενιαία αγορά να χρησιμεύει ως πρόσχημα ε, και να αντιμετωπίζονται πίσω από αυτό το παραπέτασμα, ας πούμε, οι συζητήσεις για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Θα κάνουμε ε, συζητήσεις για ποιοτικά, ποιοτικές θεραπείες που θα βασίζονται σε αποτελεσματικά φάρμακα ε, και σε φθηνά και προσιτά φαρμακευτικά προϊόντα σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων στη διάσκεψη που θα γίνει στις 6 Μαρτίου στην ε, Σόφια ε, στα πλαίσια, καθώς και μια συζήτηση στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας 22 και 23 Απριλίου. Πιστεύω ότι αυτά είναι θέματα που ενδιαφέρουν όχι μόνο τους Υπουργού Υγείας, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως συνομοθέτης, υποθέτω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται και παρακολουθεί τις προτεραιότητες, τις νομοθετικές προτεραιότητες του Συμβουλίου. Εμείς θα δώσουμε προτεραιότητα στο μοναδικό ε, νομοθετικό φάκελο που αυτή τη στιγμή είναι σε ενεργή διαδικασία, σε ενεργή φάση, στον τομέα της υγείας. Την τροποποίηση του κανονισμού για τον οργανισμό φαρμάκων, κανονισμός 726 του 2004. Οι πρώτες ε, ημερομηνίες για τους τρεμές διαλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν καθοριστεί. Αυτό το ΣΧΕ συζητήθηκε, έγιναν κάποιε πρώτε συζητήσει. Και υπάρχει περίπτωση να κλείσει αυτή η συζήτηση. Αυτό το ντοσχέ είναι τμήμα του λεγόμενου κτηνιατρικού πακέτου. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο για όλο αυτό το φάκελο και θα φτάσουμε σε συμβασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν προανήγγειλε ότι μάλλον θα υπάρξει μια νέα νομοθετική πρόταση στον τομέα Τη αξιολόγηση τη υγεία και τη τεχνολογία για την υγεία, καθώ και μια πρωτοβουλία για τα εμβόλια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η Βουλγαρία θα, θα παρουσιάσει τι προτάσει στο Συμβούλιο και θα ξεκινήσει και τη συζητήσει για αυτά τα θέματα. Όμω, θα ήθελα να τονίσω τα εξή. Για μας, η ποιότητα τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σα κάνω έκκληση λοιπόν, όσοι συμμετέχοντε στην νομοθετική διαδικασία, να συνεισφέρετε σε ένα επικοδομητικό διάλογο για τις συγκεκριμένες διατάξεις με βάση τα όσα θα γράφει το τελικό κείμενο. Το να κάνουμε μια γενική συζήτηση που θα βασίζεται σε κοινέ ιδέες δεν είναι μια αποδεκτή προσέγγιση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα αποτέλεσμα των συζητήσεων που έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να ακούσουμε τις αντιδράσει των εμπειρογνωμών των κρατών μελών, την αξιολόγηση των επιπτώσεων των εθνικών συστημάτων υγεία. Συμπερασματικά, σε όλε τι συζητήσει, το σημείο αφετηρία ε, θα είναι το να έχουμε μια καλή προοπτική για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ είναι οι συζητήσεις ζωτική σημασία για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι μπορώ να βασιστώ στην υποστήριξή σα τους επόμενου 6 μήνε. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε τον Υπουργό για άλλη μια φορά γιατί ήρθατε και για αυτή τη συζήτηση. Αρχίζουμε με το πρώτο γύρο ερωτήσεων. Δίνω το λόγο στον κύριο Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Δύο πράγματα θέλω να σχολιάσω, τα οποία παρουσιάστηκε εσείς στην παρέμβασή σας και θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά. Για, την, ε, για τον οργανισμό φαρμάκων κάναμε τη συζήτηση σήμερα το πρωί. Ε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία και θυμός για τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο έλαβε την ε, απόφαση για την έδρα της ΕΜΑ. Δεν θα κάνουμε τώρα συζήτηση επί της ουσίας, θα δεχτούμε το Άμστερνταμ, αλλά παρακαλώ να είσαστε προετοιμασμένος για το ότι το Συμβούλιο πρέπει να δώσει μια εξήγηση πώς μια τέτοια διαδικασία την οποία στο τέλος, η οποία στο τέλος ε, κατέληξε σε μια ε, κλήρωση μια τέτοια διαδικασία πώς θα γίνει να μην, να μην επαναληφθεί ποτέ. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνετε. Οι συνεργάτες σας φαντάζομαι ότι παρακολούθησαν τη συζήτηση σήμερα το πρωί, οπότε θα ήθελα αυτή τη δήλωση. Ε, προετοιμαστείτε παρακαλώ. Δεύτερον, η αξιολόγηση για την τεχνολογία υγείας. Θα ήθελα να δεσμευτείτε λίγο γι' αυτό. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η πρόταση, στις 31 ε, θα υποβληθεί και καλό θα ήταν η Προεδρία του Συμβουλίου να ξεκινήσει τη συγκεκριμένη δουλειά για τούτο το φάκελο. Σίγουρα δεν θα έχουμε στο πρώτο μισό του χρόνου συμφωνία, αλλά θα πρέπει η ομάδα εργασίας να δουλέψει επ' αυτού. Για τα κτηνιατρικά φάρμακα, σας υποστηρίζω απόλυτα. Προσπαθείτε με το Κοινοβούλιο να καταλήξετε σε μια συμφωνία. Για μας αυτό που είναι σημαντικό και δυστυχώ δεν το έχει δεχτεί το Συμβούλιο ακόμη. Εν πάση δείτε το αν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου θετικά. Στο κείμενο της Κομισιόν και του Συμβουλίου μιλάμε μόνο για τα αντιβιωτικά, τα οποία πρέπει να καταχωρούνται και να καταγράφονται. Αλλά στον ακτινιατρικό κλάδο έχουμε λιγότερα ε, ακτινιατρικά και χρειαζόμαστε λιγότερα. Αυτό δεν αναφέρεται στο κείμενο και δεν θεωρώ ότι χρειάζεται ε, να απαιτούμε μεγάλη ε, τεκμηρίωση για τα φάρμακα αυτά. Θα πρέπει να λέμε ότι θα πρέπει τα αντιβιωτικά στον κτηνιατρικό τομέα να μειωθούν. Σε ό,τι αφορά τώρα την κυρία Γκροστέτ, το Κοινοβούλιο πολλές φορές έχει ζητήσει ε, να βρεθεί μια λύση για κάποιες νέες ουσίες. Σήμερα κάθε εβδομάδα πεθαίνουν άνθρωποι είχαμε έναν ε, καθηγητή πανεπιστημιακής κλινικής ε, προσκεκλημένο και κάθε εβδομάδα μας είπε ότι πεθαίνουν άνθρωποι επειδή δεν παίρνουν τα αντιβιωτικά, δεν έχουν στη διάθεσή τους τα αντιβιωτικά που τους χρειάζονται. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει καλύτερη υγιεινή, καλύτερες, ε, καλύτερη χρήση. Χρειαζόμαστε νέες ουσίες και η Κομισιόν πρέπει σύντομα να υποβάλει πρόταση νομοθεσίας. Αυτό είναι το, η άποψη του Κοινοβουλίου. Βρίσκεται στην ε, έκθεση για τα χτινιατικά φάρμακα. Παρακαλώ, υποστηρίξτε μας, αυτή μας την, ε, σε αυτό μας το αίτημα. Πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί αλλιώς θα πεθάνουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι καθημερινά λόγω αυτού. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Στη συνέχεια ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ. Ε, στις 12 ε, πρέπει να φύγω για μία άλλη συνεδρίαση και δεν θα ακούσω τις απαντήσεις σας, αλλά θα μου τις διαβιβάσουν. Συμφωνώ με τις προτεραιότητες στον τομέα της υγείας από τη Βουλγαρική Προεδρία που είναι και προτεραιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα φάρμακα που ε, χρησιμοποιούνται για τα ζώα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μεγάλη μικροβιακή αντίσταση και φυσικά η πρώτη αιτία θανάτου είναι ο καρκίνος. Πρόκειται λοιπόν για θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν πολύ περισσότερο και βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα των αντιβιωτικών που χορηγούνται στα ζώα. Υπάρχουν ε, ολέθριες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Ναι, εντάξει, οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντιβιωτικά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και προ... περιορισμός. Και αυτό αφορά και τον μηχανισμό πάχυνσης που χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δυστυχώς ε, δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτή την ασθένεια η οποία ξεπερνάει τα σύνορα. Αυτό μας ενδιαφέρει βεβαίως είναι και η υγεία των παιδιών μας και αυτό εξαρτάται από την υγεία και την διατροφή. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη ζάχαρη και τους ε, υδατάνθρακες στα παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή για τη διατροφή των μικρών παιδιών. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ανταγωνιστικότητα της κοινωνίας μας. Τέλος, ως προς την ε, χρήση των ε, φαρμακευτικών σκευασμάτων θα ήθελα να σας πω ότι στην σχετική οδηγία θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 81 της οδηγίας του 2001 για να δούμε ποια είναι η διαδικασία προμήθειας, παρασκευής και προμήθειας των ε, σκευασμάτων. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία η πρόταση που θα υποβάλει η Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των φαρμάκων, πώς μπορούμε να ορίσουμε τις προτεραιότητες, στην έρευνα και πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα όπως θα έπρεπε. Όπως είπε ο κύριος Πέτερ Λίσε, θα πρέπει το Συμβούλιο να υποβάλει μια σοβαρή πρόταση και στόχος να είναι μια καλύτερη εργασία η συνεργασία στα πλαίσια των δικτύων και της στρατηγικής μας για να φτάσουμε σε σωστά αποτελέσματα ως προς την πρόσβαση στα φάρμακα από πλευράς πολιτών. Ο κύριος Πιέτσα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, οι προτεραιότητε της Βουλγαρική Προεδρία είναι πραγματικά ευρύτατες. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για κάποια συγκεκριμένα θέματα. Αντιμικροβιακή αντίσταση. Αυτό το θέμα γίνεται όλο και πιο σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και ένας από τους βασικούς κινδύνους για την ε, ε, δημόσια υγεία. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων παρακολουθεί την κατάσταση και οι πληροφορίες που έρχονται από το κέντρο αυτό δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε κρίση. Θα ήθελα να ρωτήσω, η Βουλγαρική Προεδρία το πρόβλημα αυτό θα το θέσει ως προτεραιότητα. Γιατί εδώ δεν μιλούμε μόνο για τους πολίτες, αλλά και για τα ζώα. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις δουλειές και για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Η αντιμικροβιακή αντίσταση και για τον τομέα αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Στην κτηνιοτροφία χρησιμοποιούνται πολύ συχνά αντιβιωτικά και για όρους πρόληψης και για την ίαση των ζώων όταν είναι ε, άρρωστα. Και υπάρχουν ε, και κάποια μηνύματα που λένε ότι παρά την απαγόρευση τα αντιβιωτικά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως ε, παράγοντες ανάπτυξης των ζώων. Υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται σχετικά και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλουμε οι εργασίες για το θέμα αυτό να ολοκληρωθούν τις επόμενους μήνες. Ε, επόμενη ερώτηση. Υπάρχουν σχέδια για την παρατήρηση των επιδημιολογικών σχεδίων για τις, ε, για τις διάφορες ασθένειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα είπαν οι συναδελφοί. Δύο πράγματα είναι σημαντικά για τη δική μας την ομάδα. Η πρόσβαση στα φάρμακα και το ερώτημά μου είναι τι μπορεί να κάνει η Προεδρία ώστε να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα και τι μπορούμε να κάνουμε και για το επιχειρησιακό μοντέλο. Θα μπορούσαμε να ε, χρησιμοποιήσουμε ένα πιο φτηνό τρόπο για να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα που τόσο απεγνωσμένα χρειαζόμαστε. Και επίσης για την ε, ομάδα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα και επαρκώς να δούμε τι γίνεται με το IMR και ποια είναι τα σχέδια της Προεδρίας, αν υπάρχουν, για την αντιμετώπιση του. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Κονέτσι να έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνουμε το ίδιο ερώτημα, νομίζω τα ίδια θέματα. Χαίρομαι που η Βουλγαρική Προεδρία μετά από ένα μισή χρόνο σιωπής θέλει να αντιμετωπίσει το θέμα των κτηνιατρικών φαρμάκων. Εμείς ε, πάντως ως Κοινοβούλιο δράσαμε πολύ γρήγορα και περιμέναμε το Συμβούλιο. Και εγώ είμαι πεπισμένη ότι η Βουλγαρική Προεδρία θα καταφέρει πολύ σημαντική πρόοδο έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και με τον τριμερή διάλογο και τουλάχιστον από την νομοθετική πλευρά η δουλειά να ε, ολοκληρωθεί. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία και χαίρομαι που το αναφέρατε κύριε Υπουργέ και εσείς. Επίσης, ο κανονισμός που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα θα μας τον αποκαλύψει η Κομισιόν. Η εντολή του Κοινοβουλίου ουσιαστικά σε λίγους μήνες τελειώνει. Οπότε θα ήθελα η Βουλγαρική Προεδρία να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της και να προσπαθήσει να κάνει όσο είναι περισσότερο δυνατά για να υπάρξει ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών, συνένεση, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον κανονισμό αυτό μέχρι το τέλος του έτους, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, τον συζητούμε χρόνια πολλά και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστεί το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο και να καταλήξουμε κάπου και χάρη στην ε, Προεδρία ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιο μονοπάτι για να επιτύχουμε τον τελικό μα στόχο. Και ελπίζω ότι δεν θα είναι μόνο σεμινάρια και διασκέψει, αλλά ότι θα βρεθεί όντω συνένεση μεταξύ των ε, κρατών μελών, έτσι ώστε και εδώ εμεί, στο Κοινοβούλιο να έχουμε μια σαφή εικόνα του πώ θα ε, προχωρήσουν τα πράγματα στο μέλλον. Ελπίζω λοιπόν ότι για τον κανονισμό που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσετε να παίξετε τον ε, ρόλο του πολύ σημαντικού ενδιαμέσου που θα βοηθήσει να ολοκληρωθεί η δουλειά φέτος. Ευχαριστώ. Ε, two more speakers. Εγώ ευχαριστώ άλλοι δύο ομιλητέ. Οπότε η κυρία Κάτεμπαχ να πάρει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας και την... τις απόψεις σας κύριε Υπουργέ. Όπως βλέπετε ένα θέμα μας ανησυχεί όλους, το θέμα της αντιμικροβιακής αντίστασης από ό,τι είδαμε και από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και θα ήθελα και εγώ να σας παρακαλέσω κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας να μπείτε εις βάθος σε αυτό το πολύ περίπλοκο θέμα. Το δεύτερο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπάρχει, υπάρχουν οι, οι θέσεις των κρατών μελών για την εφαρμογή σχεδίων δράσης, αλλά ξέρουμε ότι μέχρι στιγμής η εφαρμογή δεν έχει προχωρήσει καλά σε όλα τα κρατη Και από εκεί απορρέει και η απειλή να καταρρεύσουν τα πράγματα αν δούμε τα νοσοκομεία και την δουλειά που κάνουν και τις, ε, τα κρούσματα που αντιμετωπίζουν. Περίπου 37.000 ε, κρούσματα ε, θανατηφόρα έχουμε κάθε χρόνο στην ε, Ευρώπη αν υπήρχε κάποιος άλλος παράγων που οδηγούσε σε 37.000 θανάτους κάθε χρόνο θα το βλέπαμε πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε νομίζω το θέμα της αντιμικροβιακής αντίστασης είναι πάρα πολύ σημαντικό και προς το παρόν η εφαρμογή του δεν πάει καλά. Αυτό το One Health Approach. Αυτό το πρόβλημα θα μπορέσουμε να το λύσουμε μόνο εάν υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ των ε, υπευθύνων αρχών για την υγεία σε κάθε κράτος μέλος και για την ε, προστασία του περιβάλλοντος βεβαίω. Νομίζω ότι και εκεί από κοινού μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεύτερον, στην παρέμβασή σας, ίσως να μην κατάλαβα καλά, αλλά είπατε ότι θα πρέπει ως κοινοβούλιο τα θέματα αυτά τα, ε, της υγείας, να στα θέματα υγείας να δεχτούμε και την εθνική θέση. Το κάνουμε αυτό εφόσον βεβαίως η εθνική θέση είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας. Αλλά το άρθρο 168, 168 ε, δείχνει ποιες είναι οι αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιες είναι οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και πού μπορούμε να συνεργαστούμε. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να μπει στο προσκήνιο. Ελπίζω ότι θα το κάνει αυτό η Προεδρία, σας το περιμένω. Και ένα τρίτο σημείο θα ήθελα να ζητήσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό νομίζω, η υγιεινή διατροφή για τα παιδιά. Να μας πείτε, να μας περιγράψετε εσείς πώς στο μέλλον σχεδιάζετε να ε, διαχειριστείτε θέματα, ας πούμε, ζυζανιοκτώνων, εντομοκτώνων, ε, γλυφοσάτη, ε, γιατί μπορεί όντως να αποδεχτούν ε, ε, πολύ ε, επικίνδυνα όταν καταλήγουν στο πιάτο των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Κόβατσεφ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Να σας ευχηθώ και εγώ προσωπικά και στην ομάδα σας καλή επιτυχία. όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, η κυρία Κάντεμπαχ και οι προηγούμενοι, μίλησαν για καλή ποιοτική περίθαλψη. Και αυτό έχει να κάνει με την πρόσβαση στα φάρμακα. Με τα πιστοποιητικά, τι γίνεται για την περαιτέρω προστασία. Μιλούμε για διεύρυνση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, κυρίως όταν έχουμε ε, τα θέματα των εγκρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξέδωσε μία ε, γνωμοδότηση για το τι γίνεται σε περίπτωση άρσης για τα γενώσιμα φάρμακα. Και επίση έγινε και μία. αυτό των υποχρεώσεων για τα γενώσιμα φάρμακα. Έγινε και μία δημόσια ακρόαση και νομίζω ότι η Κομισιόν θα μα υποβάλει μία, μία πρόταση για να αλλάξει η νομοθεσία. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι η τιμή των γεννόσιμων φαρμάκων είναι πολύ πιο χαμηλή. Αν έχουμε τέτοια έγκριση για ε, πιο φθηνά φάρμακα στην αγορά, θα δούμε τη μείωση άμεσα στο κόστος και στο σύστημα υγείας και θα έχει περισσότερος κόσμος πρόσβαση στα φάρμακα, περισσότεροι ασθενείς. Οπότε εσείς ως Προεδρία τι μπορείτε να κάνετε για να μπορέσουν να υπάρξουν αυτές οι παρεκκλήσεις. Και πάλι σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία σας, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα καθήκοντά σας, ώστε ο ευρωπαϊκός πληθυσμός να έχει καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη. Ευχαριστώ. Uh, Εγώ η τελευταία ομιλήτρια, Υπουργέ. Και θα κλείσω έτσι το γύρο ερωτήσεων. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι οι προτεραιότητε της Προεδρία σας συμπεριλαμβάνουν την παιδική υγεία και ότι θα κάνετε μια διάσκεψη για την υγεία και την διατροφή για τα παιδιά. Η παιδική παχυσαρκία ε, αυξάνεται και θα φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέχρι το 2020, δεν έχουμε χρόνο. Ε, με το σχέδιο δράσης θέλουμε να περιορίσουμε την διαφήμιση α, τροφίμων σκουπιδιών για τα παιδιά και να περιορίσουμε την πρόσβασή τους ε, στα σχολεία. Η Προεδρία σας πώς θα, συμφέρει, θα συνεισφέρει σε αυτούς τους στόχους. Στην οδηγία για το οπτικοακουστικά μέσα θα υποστηρίξετε, παραδείγματος χάρη του Ροδία σας, ε, ισχυρά νομικά μέτρα για να περιορίσετε την πρόσβαση των παιδιών σε junk food. Θα δώσω τώρα το λόγο για να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι βουλευτές, να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας. Την υποστήριξη που εκφράσατε αφού ακούσατε τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας. Ακούστηκαν πολλές ερωτήσεις. Υποβλήθηκαν πολλοί άριθμα ερωτήματα, ορισμένα ε, αλληλοσπληρώνονται, ορισμένα αλληλοεπικαλύπτονται. Θα ήθελα να συνοψίσω τις ε, απαντήσεις μου, ελπίζοντας να μην ξεχνώ ότι δεν ξεχνώ καμία ερώτηση στις απαντήσεις μου. Καταρχάς, θα μιλήσω για τη διαδικασία με κατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του ΕΜΑ. Λόγω μιας απόφασης που ελήφθη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων το... στις 20 Νοεμβρίου του 2017, η Κομισιόν παρουσίασε μια πρόταση για να τροποποιηθεί ο κανονισμός του 2004-726 που αφορούσε τη μετεγκατάσταση της έδρας του ΕΜΑ από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταρτήσει μια θέση για το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο ελπίζει ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί σύντομα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να έχουμε μια συνέχεια στις εργασίες ε, του Οργανισμού Φαρμάκων. Θα σας στείλω ένα μήνυμα θα στείλω μάλλον μήνυμα στο Συμβούλιο, το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση υγεία και τεχνολογία, ή μάλλον τεχνολογική υγεία. Ε, ξέρουμε ποια είναι τα σχέδια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια νομοθετική πρόταση για την αξιολόγηση τη ε, υγειονομική τεχνολογία. Δεν την έχουμε ακόμα την πρόταση τη ε, Κομισιόν. Αλλά μια και μιλάμε για νομοθεσία, θα πρέπει να είμαστε ακριβεί. Μια και θα υπάρξει μια τέτοια νομοθετική πρόταση, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια θέματα όπως το περιεχόμενο, ο δεσμευτικός χαρακτήρας και η τελική ημερομηνία δημοσίευσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει γνώμη ε, στην αξιολόγηση αυτή στο ψήφισμα, σε ένα ψήφισμα το 2017 για τη βελτίωση ε, της πρόσβασης στα φάρμακα υπόθηκε ότι χρειαζόμαστε εθελοντική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στις προτάσεις τους. Εάν η πρόταση της Κομισιόν δημοσιευθεί, τότε η Βουλγαρική Προεδρία θα παρουσιάσει την πρόταση αυτή στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή ή στις Προπαρασκευαστικές ε, συμβουλές, ε, Επιτροπές του Συμβουλίου. Εμείς θα είμαστε ένα τίμιος διαμεσολαβητής δίνοντας αρκετό χρόνο στα κράτη-μέλη για να μελετήσουν την πρόταση και να πάρουν και να διαμορφώσουν την εθνική τους θέση. Για να προχωρήσουμε ένα φάκελο θα πρέπει να έχουμε λίγα ευαίσθητα θέματα μέσα στο φάκελο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το τελικό αποτέλεσμα αν δεν ξέρουμε, το αρχικό, αν δεν ξέρουμε και το κείμενο το τελικό. Σε ό,τι αφορά τα νομοθετικά θέματα για τη Βουλγαρική Προεδρία θα θέσουμε προτεραιότητα σε φακέλους που έχουν καλές προοπτικές να οριστικοποιηθούν. Οι προτεραιότητες μας στα φάρμακα είναι να τελειώσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το κτηνιατρικό πακέτο, πακέτο κτηνιατρικών φαρμάκων. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του κανονισμού 726 του 2004 και το κτηνιατρικό πακέτο, σε ό,τι αφορά την υγεία γενικά, προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτόν τον κανονισμό 726 που είναι και ο κανονισμός για την κατάσταση του 726 και ο κανονισμός που θεσπίζει μια κεντρική διαδικασία αδειοδότησης. Με χαρά σας αναγγέλω ότι ο πρώτος άτυπος τριμερής διάλογος έγινε στις 23 Ιανουαρίου και ήταν πολύ επικοδομητικός μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Υπάρχει συμφωνία για βασικές διατάξεις όπως ε, τέλη η υιοθέτηση τελών μάλλον και διάφορα θέματα που θα υιοθετηθούν με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Από την αξιολόγησή μα επίσης προκύπτει ότι αυτός ο φάκελος μπορεί να οριστικοποιηθεί πολύ γρήγορα. Μέσα στο πακέτο υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, όπως μικροβιακή αντοχή. Πιστεύουμε ότι οι συνομοθέτες ενδιαφέρονται να βρεθεί μια καλή λύση προς το συμφέρον της υγείας και ελπίζω αυτό να συμβεί για όλο το πακέτο. Σε ό,τι αφορά τη μικροβιακή αντοχή, η μικροβιακή αντοχή αναγνωρίζεται ως σημαντικό θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σοβαρή η πρόκληση και απειλή για την υγεία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015 υιοθέτησε ένα ψήφισμα για μια ασφαλή υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής και βελτίωση της προστασίας υγείας των ασθενών. Το 2016 υιοθετήθηκαν συμπεράσματα από το Συμβούλιο για τα επόμενα βήματα στα πλαίσια της προσέγγισης για την ενιαία υγεία. Αυτό το σχέδιο ενιαία υγεία που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2017 από την Κομισιόν θα οδηγήσει τώρα σε μια εθνική εφαρμογή του. Κάθε κράτος μέλος έχει τα δικά του μέτρα εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, περιστάσεις στην επικράτειά του. Εμείς έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες ε, για να εφαρμόσουμε ένα εθνικό σχέδιο καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής. Σε ό,τι αφορά τι νομοθετικέ λύσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα πλαίσια του κτηνιατρικού πακέτου, υπάρχουν σημαντικές πτυχέ που συνδέονται με τη μικροβιακή αντοχή. Επομένω ω Προεδρία, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ληφθεί μια απόφαση με βάση αυτή την προσέγγιση ενιαία υγεία. Η ενιαία προσέγγιση για την υγεία. Ε, έχουμε μια έκθεση της, ε, του ΕΜΑ για την, ε, τις πωλήσει και τη χρήση. Τώρα, για την υγιεινή διατροφή των παιδιών. Ένα από τα οριζόντια θέματα είναι το θέμα των νέων και των παιδιών και που είναι η καλύτερη επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης και βεβαίως για να είναι καλή αυτή η επένδυση θα πρέπει να είναι υγιή τα παιδιά. Ε, αν υγιή τα παιδιά και οι νέοι σημαίνει παραγωγική, ε, παραγωγικό εργατικό δυναμικό αυτό συνδέεται με πρωτοβουλίες που έχουν προωθήσει άλλες προεδρίες και συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η ελληνική, η ολλανδική και η μαλτέζικη προεδρία έχουν υιοθετήσει σχετικά συμπεράσματα. Με χαρά βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει προτεραιότητα σε αυτό το θέμα και κυρίως στο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση παχυσαρκίας των παιδιών. Κάνουμε όμως αρκετά για να δώσουμε ένα ε, υγιεινό μοντέλο στα παιδιά και μια υγιεινή διατροφή. Η διατροφή είναι μία από τις βασικές πτυχές που εξασφαλίζει καλή υγεία. Ε, έχουμε απίστευτη άνοδο των χρόνιων ασθενειών που απορρέει και τον τρόπο που τρώμε. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό ε, και εστιάζουμε εδώ στην υγεία. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το θέμα της υγείας και να την εφαρμόσουμε σε όλες τις πολιτικές. Ε, η διατροφή και τα ποιοτικά τρόφιμα θα πρέπει να μας βοηθήσουν τόσο ώστε να έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μέτρα προφύλαξης και προληπτικές πολιτικές. Επομένως, τα τρόφιμα μπορούμε να τα δούμε από διάφορες πτυχές. Έχουμε να κάνουμε την απασχόληση, εμπόριο, περιβαλλοντική προστασία, επιστήμη, ανάπτυξη, έρευνα. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η επίπτωσή του στην ανθρώπινη υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία. Έγιναν συζητήσει για την ανάγκη για τρόφιμα, όχι μόνο ασφαλή, αλλά και υγιεινά. Μιλάμε για την παραγωγή που θα πρέπει να βασίζεται σε υγιεινά, στην, στην ιδέα ότι πρέπει να παράγονται υγιεινά τρόφιμα, όχι μόνο στις απαιτήσει του καταναλωτή, στη ζήτηση. Ε, επίσης θα συζητήσουμε και την επίπτωσή τους ε, στην υγεία των παιδιών, καθώς και το ρόλο των παραδοσιακών μοντέλων διατροφής στην Ευρώπη και την επίδρασή τους στην υγεία, την ανάγκη να διατηρήσουμε την, μια ποικιλομορφία ε, στα τρόφιμα. Τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα είναι οι πιο ευάλωτοι καταναλωτέ, δεν μπορούν να κάνουν υγιεινέ επιλογέ από μόνα του. Γι' αυτό ε, σε αυτή την προτεραιότητα, η κοινή διατροφή για τα παιδιά, ετοιμάζουμε μία ε, διάσκεψη σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων που θα γίνει στη Σόφια στις 6 Φεβρουαρίου και θα υπάρξουν και συμπεράσματα εν συνεχεία του Συμβουλίου. Η υγεία στη... και η γεωργία είναι δύο πράγματα που πρέπει να πορεύονται μαζί. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει πολιτική συνένεση για το θέμα αυτό. Ο στόχος μας είναι να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, πώς μπορούμε να έχουμε συντονισμό για θέματα ε, υγείας και γεωργίας, ούτως ώστε να παράγουμε υγιεινά τρόφιμα. Αυτό συνδέεται επίσης με την αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Οι πτυχές της υγείας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και σε αυτό το επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα, θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις που αφορούν τα φάρμακα. Γιατί είναι περίπλοκο το θέμα και είναι τμήμα των προτεραιοτήτων της, προτεραι... Μία από τις προτεραιότητες ακριβώς είναι η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Αποτελεσματικότητα, θεραπευτικός πώς, αλλά και να υπάρχει καλή σχέση κόστους-οφέλους, ε, το... η επίπτωση που έχουν στο σύστημα υγείας και η αποτελεσματικότητά του. Ε, το να μην υπάρχουν ε, φάρμακα γιατί είναι πολύ ακριβά ή γιατί δεν είναι αρκετά, ε, καθώς και το θέμα των εξαγωγών είναι βασικά στοιχεία τη συζήτηση, καθώ και η επίπτωση στον προπολογισμό των κρατών μελών, επίπτωση του κόστου των φαρμάκων. Οι συζητήσει για αυτά τα θέματα έγιναν ε, επί σειρά προεδριών, στην Ελληνική Προεδρία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, ε, Ολλανδία, ε, Σλοβακία και Μάλτα. Σε όλε αυτέ τι προεδρίε έγιναν τέτοιε συζητήσει. Μια σημαντική συνεισφορά στη συζήτηση γίνεται και από τα όσα λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υιοθετήσατε το 2017 ένα ψήφισμα για τη βελτίωση τη πρόσβαση ε, στα φάρμακα. Ε, οι τιμέ λοιπόν των φαρμάκων, η θε, θεραπευτική του επίπτωση, η οικονομική κατάσταση των κρατών μελών, όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν μιλάμε για την πρόσβαση στα φάρμακα. Αυτέ οι συζητήσει θα πρέπει να είναι τμήμα της ατζέντα του Συμβουλίου, ούτως ώστε να βρεθούν πιθανές λύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω κάποια βασικά θέματα σε αυτό το τομέα. Η έλλειψη φαρμακευτικών σκευασμάτων σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι που, κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Γιατί ε, όπως γνωρίζετε, το θέμα των φαρμάκων δεν είναι απλό. και αυτό χρειάζεται μία συζήτηση για την διάθεσή του στην αγορά. Η Βουλγαρία έχει αναλάβει μέτρα για να ανοιχνεύσει αυτή την ανεπάρκεια φαρμάκων έχουμε προβεί στη σύσταση ενός ηλεκτρονικού συστήματος σε σχέση με την διάθεση και πληρωμή από δημόσιο χρήμα των φαρμάκων και θα υπάρξουν και κυρώσεις εκεί που θα χρειαστεί. Επίσης, ως προς την διαπραγμάτευση των τιμών των φαρμάκων, θα πρέπει να δούμε ορισμένα περιφερειακά συμβατικά ζητήματα και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια της τιμολόγησης. Χρειάζεται αυτή η διαφάνεια για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε στο τέλος τέλος να υποστηρίξουμε τους ασθενείς. Αυτό είναι και το απότερο μέλημά μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν δίκαιο ανταγωνισμό για να λειτουργήσει καλά η αγορά και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ μεγάλες εξουσίες για την προστασία του ανταγωνισμού. Άρα θα πρέπει να προωθηθούν πρωτοβουλίες από την Επιτροπή και το Συμβούλιο περιμένει και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πνευματικά δικαιώματα. Η Βουλγαρική Προεδρία θέλει να οργανώσει μια διάσκεψη εμπειρογνωμόνων στις 6 Μαρτίου το 2018 στη Σόφια για να ασχοληθούμε με το τρέχον ζήτημα καθώς και στο Συμβούλιο Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ένας δελεαστικός χώρος για την παρασκευή φαρμάκων. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για την γλυφοσάτη. Το ζήτημα αυτό έχει συζητηθεί σε επιτροπές εργασίας ως προς την γεωργία, αλλά υπάρχουν και πτυχές που άπτονται της υγείας. Όπως ξέρετε η Επιτροπή ανέλαβε μία εκτελεστική πράξη για την ανανέωση της χρήσης της γλυφοσάτης μετά από σοβαρές συζητήσεις μεταξύ κρατών μελών και έγινε λόγος για μια πενταετή περίοδο βαθμίας απαλυφής της ε, γλυφοσάτης. Η Επιτροπή λοιπόν θα μας ενημερώσει έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια για αυτό το phasing out και να δούμε ποια βήματα θα ακολουθήσει και η ΕΦΣΑ. Τέλος, ως προς την άρση της πιστοποίησης προϊόντων προστασίας, ε, όπως γνωρίζετε ως προς τα γενώσιμα, η Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα δελεαστικός ε, χώρος για την παρασκευή αυτών των φαρμάκων. Άρα θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις, διότι θα πρέπει να παράγουμε γενώσιμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί εξαρτόμαστε από παρασκευαστές από τρίτες χώρες, κάτι το οποίο δεν είναι υπέρ του συμφέροντος των ασθενών ή τη γενικότερη υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα γίνεται μία δημόσια διαβούλευση σε σχέση με αυτή την άρση της πιστοποίησης. Μιλάμε για ένα 10 συν 5 προστασία τεχνίας. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η καταλεκτική ημερομηνία, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μία απάντηση και σε αυτό το θέμα των γενοσύμων. Εάν ε, συζητηθεί αυτό το θέμα επί Προεδρίας μας, θα το συζητήσουμε στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό γιατί ε, απάντησε σε πληθώρα ερωτήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί μας παρουσιάσατε τις ε, προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Είδα ότι συμμεριζόμαστε πολλές από αυτές τις προτεραιότητες, τις προτεραιότητες και γι' αυτό εξ ονόματος όλων των Ευρωβουλευτών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент, за мен бе Ευχαριστώ που και εγώ με τη σειρά μου ήταν ε, μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Νομίζω ότι χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ύψης της σημασίας και ως Προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να έχουμε πολύ καλή συνεργασία και επικοινωνία, να χρησιμοποιήσω τις καλές πρακτικές που προϋπάρχουν και σε υψηλότερο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. This was uh, the last point, so bon appetit.